Okay, good afternoon everybody. Welcome to this sitting of the committee and um, I call the committee to order. Καλημέρα σας. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε είμαι απλώς ο γυρεότερος τη τάξη διότι απουσιάζει και η πρόεδρος και η αντιπρόεδρη αυτή τη στιγμή. Το πρώτο θέμα στην μερίσια διάταξη λοιπόν είναι η έγκρισή τη. Υπάρχει κάποιο ο οποίο θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο για την ημερήσια διάταξη. Η σιωπή σα σημαίνει ότι συνενείται, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Και το επόμενο σημείο είναι οι ανακοινώσει του Προέδρου. Μία ανακοίνωση. Να σας επιβεβαιώσω ότι υπάρχει διερμηνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες σήμερα. Αύριο θα λείπει μία γλώσσα και θα σας πει η πρόεδρος ε, αύριο. Σε ποια γλώσσα δεν θα μπορείτε να μιλήσετε και να ακούσετε. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να περάσουμε. Δεν έχουμε τίποτα να εγκρίνουμε από πρακτικά. Στο πρώτο σημείο της ημερήσια διάταξη λοιπόν έχουμε την κοινή συζήτηση για τον ορίζοντα 2020. Θα το συζητήσουμε ανατμήματα το ζήτημα. Το πρώτο τμήμα θα είναι η έκθεση της κυρίας Ρέιρα Μαντουρέλ. Στη συνέχεια θα μιλήσει κυρία Καρβάγιο. Θα κάνουμε, θα ακούσουμε λοιπόν δύο εναρκτήριες ομιλίες. Ε, στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους και σας ε, ενημερώνω ότι θα προσπαθήσω να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και αν καθυστερήσετε πάνω από δύο λεπτά θα σας διακόπτω. Ε, στη διακριτική ευχαίρεια του Προέδρου βέβαια αυτό. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση λοιπόν, αν η κυρία Ρέιρα Μαντουρέλη είναι έτοιμη να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, το να σας βλέπω στο Προεδρείο μου θυμίζει παλιούς καιρούς και όπως είπατε και εσείς δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Ε, ας επιτρέψτε μου λοιπόν να σας εξηγήσω κάποιους από τους ε, λόγους, ε, οκτώ έχω επιλέξει, που μας οδήγησαν στο να καταθέσουμε τις τροπολογίες τις οποίες έχετε αναχείρας, τροπολογίες στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο πρώτος λόγος ήταν καταρχάς να αντιμετωπίσουμε την κρίση για να ξεφύγουμε από την παρούσα κρίση και να ε, αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τοποθετηθεί σαφέστατα στην οικονομία της γνώσης. Αυτό είναι το πλαίσιο που καθορίζει τη στρατηγική της Ευρώπης 2020 και θα μπορέσει να είναι επιτυχές μόνον εάν ε, ε, διατηρήσουμε τη σταθερότητα του συστήματος έρευνας και ανάπτυξης και σε οικονομικούς αλλά και σε ανθρώπινους πόρους. Και είναι απολύτως απαραίτητο στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020 να υπάρχει διπλάσιος προπολογισμό σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο το οποίο είναι ενισχύει αυτή τη στιγμή. Η δεύτερη μεταβλητή από την οποία ε, ε, εξαρτάται αυτή η διαδικασία είναι οι ανθρώπινοι πόροι. Χωρίς επιστήμονες και ερευνητέ, δεν υπάρχει έρευνα και δεν υπάρχει καινοτομία πάνω στην οποία θα πρέπει να οικοδομηθεί η οικονομική ανάπτυξη την οποία επιθυμούμε. Γι' αυτό και ακριβώς στην έκθεση έχουμε καταθέσει μια σειρά από τροπολογίες που στόχο έχουν να ενισχύσουν τη δυνατότητα να προσελκύσουμε, να διατηρήσουμε αλλά και να προωθήσουμε τα καλύτερα ταλέντα και ε, έχουμε ζητήσει να ειθαχθούν και δείκτες για τους ανθρώπινους πόρους ως αναπόσπαστο τμήμα της αξιολόγησης του ορίζοντα 2020. Ο δεύτερος από τους λόγους είναι να εγγυηθούμε πραγματικά τη συνέχεια της αλυσίδας της καινοτομίας να ενσωματώσουμε ε, στις ε, ερευνητικές δραστηριότητες την ε, καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την νέα αρχιτεκτονική του προγράμματος και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε να έχουμε ισορροπία μεταξύ των διαφόρων ε, πτυχών της αλυσίδα. Δηλαδή, κατά βάση την έρευνα και την καινοτομία, ιδίω σε όρους προπολογισμού. Εξίσου σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι θα ενσωματωθούν ε, τα διάφορα στάδια της καινοτομία. Γι' αυτό στην έκθεση θεωρούμε ότι πρέπει να βελτιωθεί ε, η δημιουργία ενός δικτύου των τομεακών διευθυντικών ομάδων και δημιουργείται και ένα τμήμα ε, κάτω από το μηχανισμό κεφαλαίου. Ο τρίτος λόγος είναι φυσικά η εμπιστοσύνη στην αριστεία. Θα πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο αριστείας της επιστημονικής βάσης της Ευρώπης και να θεμελιώσουμε τα επιστημονικά ταλέντα του αύριο. Αυτό κατά την άποψή μου δικαιολογεί απολύτως ε, το γεγονός ότι ο πυλώνας ε, για την αριστεία θα πρέπει να λαμβάνει το 1 τρίτο της χρηματοδότησης του προγράμματος. Τέταρτον, να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες ε, προκλήσεις. Εδώ, σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, ο στόχος ενέργεια ε, αυξάνεται σημαντικά στον προπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ζήτησε αυτό επανειλημμένο σε αρκετά ψηφίσματα. Επιπλέον, υποστηρίζουμε τους στόχους της μείωσης διοξιδίου του άνθρακα, τους οποίους υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε τα δύο τρίτα της χρηματοδότησης που προβλέπονται για την ενέργεια να ε, αφιερωθούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλω να σας πω επίσης ότι η έκθεση για την προτεραιότητα 3 για τις κοινωνικές προκλήσεις διατηρεί κατά βάση την δομή που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εξαίρεση τις ε, κοινωνίες που περιλαμβάνουν τους πάντες, ε, το οποίο έχει διαιρεθεί σε δύο τμήματα. Αφενός έχουμε την πρόκληση του να καταλάβουμε τις ε, κοινωνικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης να προστατεύσουμε την ελευθερία και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Κατά αυτόν τον τρόπο οι κοινωνικές επιστήμες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες για το πρώτο τμήμα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όταν θέλουμε να προχωρήσουμε σε κοινωνίες που θα περιλαμβάνουν τους πάντες και θα είναι πιο καινοτόμες. Με τις τροπολογίες αυτές θέλουμε, και αυτό ε, είναι και το πέμπτο αίτιο το οποίο θα σας αναφέρω, να ενισχύσουμε το διαρθρωτικό χαρακτήρα του προγράμματος πλαίσιο ορίζοντας 2020. Τα προηγούμενα προγράμματα πλαίσιο διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο διαρθρώθηκε το σύστημα της τεχνολογίας και των επιστημών στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της χρηματοδότησης ε, δράσεων που μας ε, βοήθησαν να προωθήσουμε εξαίρετους επιστήμονες και εξαίρετες ιδέες. Και εδώ ε, ο στόχος στην έκθεση είναι να προστατεύσουμε αυτό το ε, κτήμα που έχουμε αποκτήσει και να προσπαθήσουμε να έχουμε δράσεις οι οποίες θα είναι υπέρ της ανταγωνιστικότητας και σε ε, όλους τους τομείς να μπορέσουμε να έχουμε χρηματοδότηση για μεγάλα προγράμματα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν και στη συμμετοχή νέων συμμετοχόντων και να δώσουν το δέοντα ρεολισμό στο σύστημα. Γι' αυτό ακριβώς αυξήθηκε και η χρηματοδότηση των δράσεων Marie Curie και των ερευνητικών ιδρυμάτων. Ε, δίνουμε ιδιαίτερη, ιδιαίτερη σημασία στις infrastructures και επίσης έχουμε και ένα νέο συγκεκριμένο στόχο να επεκτείνουμε την αριστεία για να διευρύνουμε τη συμμετοχή με στόχο να ενισχύσουμε τον επιστημονικό ιστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, έχω τρία ακόμα σημαντικά αίτια. Ε, θα τα αφήσω για τη συζήτηση, αλλά επιτρέψτε μου να μιλήσω λιγάκι ακόμα, διότι δεν θα ήθελα να ολοκληρώσω χωρίς να ευχαριστήσω. Ο πρόεδρος Διακόπτη θα σας δώσω λίγο περισσότερο χρόνο αν υπάρχει στο τέλος και θα μας πείτε τα τρία σημαντικά σημεία. Ένα λεπτάκι μόνο για να ευχαριστήσω τη γραμματεία τη Επιτροπής μα, τη γραμματεία τη ομάδα μου, το γραφείο μου για όλη τη βοήθεια που μου έδωσαν για να ετοιμάσω αυτή την έκθεση. Να ευχαριστήσω και τους κοιόδη συζητητέ από τι διάφορε ομάδε και του συζητητέ από τι υπόλοιπε εκθέσει ε, που όλοι μαζί έχουμε όλο αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε και για τι εντατικέ συζητήσει που κάναμε, για τη βοήθειά σα και για τη διάθεση να καταλήξουμε σε συμφωνία ε, να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αγαστή συνεργασία και το Συμβούλιο. Ε, η Ιδανική Προεδρία μας βοήθησε ιδιαίτερα. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα και με τη βοήθεια της συνεργασία όλων ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι είχε συμφωνηθεί ο χρόνος αγόρευσης. Εν πάση περιπτώσει χαίρομαι γιατί καταφέρατε να πείτε όσα θέλατε σε αυτό το χρόνο, αλλά θα είμαι πολύ πιο αυστηρό μετά. Η κυρία Καρβάγιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω του συναδέλφου έτσι ώστε να μην ε, ξεχαστώ και να μην με κόψει ο Πρόεδρος στο τέλος ε, του εισηγητές των άλλων ε, εκθέσεων, τους σκιώδησε και την καλή συνεργασία με το Συμβούλιο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά τον ορίζοντα 2020 και αναφέρει ε, προτεραιότητες. Επομένως, ε, συνεχίζουμε από εκεί που ε, σταματάει η έκθεση της κυρίας Ριέρα Μαντουρέλ. Τέσσερα είναι τα κύρια στοιχεία της έκθεσής μου. Πρώτον, η αριστεία Όσον αφορά την αριστεία, αυτό θα πρέπει να είναι το κύριο στοιχείο του ορίζοντα 2020. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι θα υπάρχει διεύρυνση της συμμετοχής έτσι ώστε να υπάρχει όθηση της αριστείας σε ολόκληρη την Ευρώπη και έτσι να υπάρχει επιστημονική αριστεία bottom-up σχετικά με τον ορίζοντα 2020. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή την κλίμακα ε, προς την αριστεία. Κατά την έννοια αυτή έχω υποβάλει πολλές τροπολογίες έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η stairway to excellence, αυτή η κλίμακα προς την ε, ε, αριστεία. Το δεύτερο σημείο μου είναι η οικοδόμηση συνεργειών μεταξύ του ορίζοντα 2020 και των διευθυντικών ταμείων. Έχουν συμπεριληφθεί στοιχεία στην έκθεση, στόχος των οποίων είναι η δημιουργία καλύτερης συνέργειας μεταξύ των δύο προγράμματων. Επίσης, ε, το ε, ας πούμε στοιχεία όπως είναι η ε, ετικέτα της αριστείας σε καλά προγράμματα, ο συν, η συγχρηματοδότηση όσον αφορά τα διάφορα πιλωτικά προγράμματα και τα προγράμματα επίδειξης ε, θεωρούμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί ε, μια καλή συνέργεια και με την κοινωνική διάσταση. Ε, επίσης, θέλουμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Δεν θα πρέπει να έχουμε μείωση της συμμετοχής. Αντιθέτως, ε, θα πρέπει τα ευρωπαϊκά προγράμματα και η συμμετοχή να αφορά και τους τρεις πυλώνες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βεβαίως θα πρέπει να ε, συμμετέχουν και κατά αυτή την έννοια έχω υποβάλει πολλές ε, τροπολογίες. Ας πούμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε και ένα σύστημα δελτίου καινοτομία, Innovation Voucher. Οριζόντια θέματα επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται Ήδη κάποια οριζόντια θέματα έχουν ε, υπογραμμιστεί. Ε, ας πούμε τα θέματα σε σχέση με τον ορίζοντα 2020 καθώς επίσης και ο διάλογος μεταξύ κοινωνίας ε, και και επιστημόνων, καθώς επίσης και η επίλυση κάποιων οριζοντίων προβλημάτων. Κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τις πρωτοβουλίες οι οποίες ήδη περιέχονται στην πρόταση της Κομισιόν, ε, πρέπει να πω ότι εγώ έχω υπογραμμίσει κάποια σημεία τα οποία είναι ιδιαίτερης σημασίας ε, και τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί όπως θα έπρεπε με την απαραίτητη έμφαση. Το νερό, το φυσικό αέριο, ε, η πολιτιστική κληρονομιά, η αποθεματοποίηση της ενέργειας. Πριν ολοκληρώσω θα ήθελα να επανέλθω στο γεγονός ότι ε, στην έκθεσή μου προσπαθώ να ευθυγραμμιστώ και με την έκθεση της κυρίας Μαντουρέλ. Επίσης να πω ότι επέλεξα ε, στο πλαίσιο της ε, κοινωνικής πρόκλησης υπαριθμών 6 ε, επέλεξα να διατηρήσω τη σχέση μεταξύ κοινωνίας και επιστήμης. Εν είδη συμπεράσματος να σας πω ότι θα ήθελα να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων και με μεγάλη χαρά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 εκπροσωπώ βεβαίως ε, τη, τον ε, κανονικό σκιώδη. Θα είναι όμως ε, εδώ για αύριο, δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας. Και έχω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Μαδουρέλε για την εξαιρετική έκθεση η οποία αντιμετωπίζει πολλά σημαντικά θέματα και τα οποία μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση για τις επερχόμενες συζητήσεις. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την κυρία Μαδουρέλ για την επικοδομητική της στάση και την καλή συνεργασία. Τους τελευταίους μήνες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέπτυξε μια συνεκτική ε, και ισχυρή θέση απέναντι στον ορίζοντα 2020. Ακόμα περισσότερο όμως και πιο σημαντικό αναπτύξαμε τον θεμελιώδη ρόλο που θα πρέπει να παίξουμε σε σχέση με την καινοτομία και το ρόλο που θα πρέπει να παίξει η καινοτομία ε, στο μέλλον της ε, Ευρώπης. Είναι σαφής οι προτάσεις της κυρίας Μαδουρέλ για τον ορίζοντα 2020 ε, και ο χρηματικός στόχος των 100 δις ευρώ. Ε, έχουμε ε, έξι στόχους και πιστεύουμε ότι ε, το υπόβαθρο το οποίο οδήγησε στους έξι αυτούς στόχους έχει καλυφθεί πλήρως. Είναι γνωστό αυτές ε, οι οικονομικές ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζει τώρα η Ευρώπη και επομένως ε, θα πρέπει με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπίσει αυτά τα σημεία τα οποία αναφέρονται στην έκθεση. Θέλουμε αριστεία και μάλιστα διευρυμένη αριστεία στον ορίζοντα 2020 και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μια σημαντική δουλειά που έχουμε μπροστά μας. Ο ορίζον 2020 οπωσδήποτε θα πρέπει να παράσχει τα απαραίτητα εργαλεία έτσι ώστε να δώσει στην καινοτομία και στην επιστημονική αριστεία τις θέσεις που τους αρμόζουν. Ε, θα πρέπει να ε, δοθεί στην ερευνητική ε, κοινότητα κάθε δυνατότητα έτσι ώστε να μπορέσουν να παίξουν το ρόλο που τους αρμόζει. Όλα αυτά τα οποία αναφέρει η κυρία Μαδουρέλη σε σχέση με τον ορίζοντα 2020 2020 θα πρέπει να στηριχτούν. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Είναι, αυτά μου έχει γράψει ο συνάδελφος, πρέπει να τα τελειώσω. Ε, όσον αφορά ε, την ε, Όσον αφορά το χώρο έρευνας και ασφάλειας, ε, πολλά θα πρέπει να γίνουν ακόμα. Ε, έχω και άλλα στοιχεία εδώ, κύριε Πρόεδρε, αλλά φαίνεται δεν έχω το χρόνο να τα αναφέρω. Ε, νομίζω να σταματήσω εδώ και ενδεχομένως να κάνω κάποια άλλα σχόλια αργότερα. Τέλος, τέλος, να πω την τελευταία φράση. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να βάλει τον ορίζοντα 2020 στη θέση που του αρμόζει και αυτό θα πρέπει να είναι το κεντρικό στοιχείο των ε, συζητήσεων που γίνονται για την οικονομική ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ίσως αργότερα, λέει ο Πρόεδρος, να έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε κάποια πράγματα. Η κυρία Χόλ τώρα. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω εκ μέρους του Μακένζι Χάνσον, του οποίου έχει καθυστερήσει η πτήση δυστυχώς. Καταρχά να ευχαριστήσω του συζητητές για τις εκθέσει τους και θα ήθελα να κάνω τρει με τέσσερι παρατηρήσεις. Το Horizon 2020 δεν είναι απλό το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, δεν αφορά μόνο την έρευνα αλλά και την καινοτομία. Ο κύριος Χάνσον λοιπόν ανησυχεί λίγο διότι υπάρχει μια τάση να επικεντρωθούμε ε, σε άλλες δραστηριότητες και όχι σε δραστηριότητες που είναι πιο κοντά στις αγορές και να ε, επικεντρωθούμε περισσότερο στη βασική έρευνα. Η βασική έρευνα είναι και αυτή σημαντική και τα δύο είναι αναπόσπαστα τμήματα ενός συνόλου και πρέπει να έχουμε αυτή την προσέγγιση. Ε, επίσης, ε, η πρόταση του Συμβουλίου, η προκλήση για την κοινωνία, δηλαδή από έξι να γίνουν δύο και να δώσουμε και ιδιαίτερα έμφαση στην ασφάλεια, ο ε, σκιώδης ε, των φιλελευθέρων θεωρεί ότι αυτό ο διαχωρισμός είναι δυστυχής, διότι θα χαθεί το σημαντικό στοιχείο των κοινωνικών επιστημών ε, στην κοινωνική ασφάλεια. Και είδαμε ότι μετά τη Φουκουσίμα, ότι μετά από τις πλημμύρες και τα θέματα της αλλαγής του κλίματος, υπάρχει και μια περιβολητική πτυχή που άπτεται τη ασφάλεια. Εάν λοιπόν διαχωρίσουμε αυτούς του τομεί. ε, το περιβαλλοντικό και το ανθρώπινο στοιχείο μπορεί να χαθούν και να μείνουμε μόνο στην τεχνολογία. Τρίτον, ο σκιώδης ηγητής των φιλελευθέρων συμφωνεί με την αρχή η οποία διέπει το προτινόμενο 50% ε, της ανάθεσης συγκεκριμένου προπολογισμού, αλλά θα ήθελα να συζητηθεί λίγο αυτό το ποσοστό. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι να υπάρχει ένα πρόγραμμα πλαίσιο το οποίο θα είναι απλουστευμένο και θα τους διευκολύνει τη συμμετοχή. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι αναγνωρίζει τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διαδικασία, δεν είναι απόλυτα πεπισμένο ότι το να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό στον προπολογισμό για αυτούς είναι η σωστή απάντηση. Και τέλος, ε, χαιρετίζω προσωπικό στην αναφορά που γίνεται στην αναφορά του ε, τα δύο τρίτα του προπολογισμού της ενέργειας να πάνε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βλέπουμε την πρόταση για το 2050 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και καλό θα ήταν να γίνει έρευνα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα πρέπει να την υποστηρίξουμε χρηματοδοτικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Φόρτ στη συνέχεια. Για δύο λεπτάκια περίπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τις δύο εισηγήτριες. Έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και όλους τις ηγητές για τον τρόπο με τον οποίο έκαναν συνεδριάσεις και συμπεριλάμβαναν τους πάντες ε, μέχρι σήμερα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να σταθώ σε τρεις πτυχές. Την αριστεία, τα ποσοστά χρηματοδότησης και την ανοιχτή πρόσβαση ως προτεραιότητα. Στόχο είναι να χρηματοδοτήσουμε την καλύτερη έρευνα και την καλύτερη καινοτομία στην Ευρώπη. Ε, το θέμα τη ευρύτερη συμμετοχή λοιπόν είναι σημαντικό, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να είναι ει βάρο της επιστημονικής αριστείας. Και ξέρω ότι και οι δύο έχετε βάλει νέου τίτλου και θέλετε να έχουμε μεγαλύτερη αριστεία και να διευρύνουμε τη συμμετοχή. Εγώ προτιμώ την προσέγγιση τη κυρία Καρβάγιο ε, να βρίσκονται τα πάντα εντό του προγράμματο ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ταμεία συνοχή σε άλλους ε, ε, πόρους ε, με συνέργειες που θα μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους όπως τους επιθυμάτε. Η κυρία Μαντουρέλ λέει ότι θα πρέπει να διευρύνουμε τη συμμετοχή στον πυλώνα της αριστείας. Ίσως αυτή η πρόταση μπορεί να είναι εις βάρος της αριστείας και νομίζω ότι αυτό δεν είναι προ όφελο κανενό. Καλό θα ήταν λοιπόν να γίνει με συντονισμό μεταξύ των διαφόρων πτυχών. Τώρα, για τη χρηματοδότηση εν γέννη από τους ενδιαφερομένους με τους οποίους συναντήθηκα, ο καθένα ζητάει περισσότερα χρήματα και θέλει να αναφέρεται ο τομέας του. Νομίζω ότι θα πρέπει ή δυνατόν να υπάρχει μια κάποια ευελιξία, διότι όπως γνωρίζουμε προκύπτουν νέε προκλήσεις ε, και θα προκύψουν και στο μέλλον και αυτό που γνωρίζουμε σήμερα μπορεί να μην είναι η πραγματικότητα του 2018. Καλό είναι λοιπόν να υπάρχει μια κάποια ευελιξία. Όσον αφορά το θέμα της μεγαλύτερης συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εγώ ανέκαθεν έλεγα ότι αυτό επιτυγχάνεται μέσω απλούστευσης. Να επισημάνω όμως ότι ε, από αρκετά κράτη-μέλη υπάρχουν αιτήματα ε, για περισσότερη και ζητείτε να υπάρχουν περισσότερα προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε. Ίσως λοιπόν ε, θα έπρεπε εν μέρη να έχουμε απλούστευση και εν μέρη να στοχεύσουμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να το επιτύχουμε. Όσον αφορά την ανοιχτή πρόσβαση, υποστηρίζω την αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, ιδίως σε κάποιους τομείς της επιστήμης, αλλά θα πρέπει να γίνει με βιώσιμο τρόπο, χωρίς να περιορίσουμε τα επιχειρηματικά μοντέλα ε, και τη δημοσίευση των εργασιών, διότι αυτή είναι προστιθέμενη αξία για την επιστήμη. Το κόστος λοιπόν της δημοσίευσης θα πρέπει να καλύπτεται από κάπου αλλού. Εάν δεν πληρώνετε λοιπόν να διαβάσετε θα πρέπει να βοηθήσουμε ε, ε να καλύπτεται το κόστος εκτύπωσης. Η κυρία Μαντουρέλ πρότεινε ε, να υπάρχουν αρκετές διευθυντικές ομάδες. Όλοι θέλουμε να υπάρχει χρηστή διακυβέρνηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Θα πρέπει να το επεξεργαστούμε περισσότερο. Όσον αφορά την ισότητα των φέλων, ε, θέλουμε να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες σε υψηλές θέσεις, αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει ένα άρθρο που να αναφέρεται σε αυτό και όχι να είναι διάσπαρτο με στο κείμενο. Να διασφαλίσουμε ότι και οι γυναίκες και οι άνδρες που επιστρέφουν στο χώρο μετά από κάποια διακοπή, κάτι το οποίο είναι σύνηθες, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε και γυναίκες στο χώρο αριστείας. Ευχαριστώ. Κυρία Ματία, και εσεί αναφέρεστε ω κοιόδη εισηγήτρια και ξέρω ότι θα μιλήσετε ω εισηγήτρια στο επόμενο. Θέλετε να πείτε κάτι για το θέμα αυτό. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ναι, ευχαριστώ πολύ σύντομα. Και εγώ θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντα του συναδέλφου για τη δουλειά που έκαναν. Εμείς ε, Έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτές τις δύο εκθέσεις που προφανώς είναι ευδιάκριτο ότι υπάρχει μεγάλη συνδιάρθρωση, συνάρθρωση μεταξύ αυτών των δύο εκθέσεων. Υπάρχουν μικρές διαφορές αλλά έγινε μεγάλη δουλειά από κοινού εδώ. Κυρίως θέλω να υπογραμμίσω κάποια θέματα. Θέλω να ενισχύσω κάποια άλλα όσον αφορά την υποστήριξη για τις προτάσεις που μας παρουσιάζονται εδώ. Και για, στις γενικές γραμμές οι δύο εισηγήτριες, οι δύο εισηγήσει καταφέρνουν να παρουσιάσουν μια πρόταση που επιτρέπει να τοποθετήσουμε αυτό που είναι ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα όπως η έρευνα και η ανάπτυξη στο επίκεντρο και να δώσουμε πρόσθετη αξία ακριβώς σε μια κατάσταση που έκδηλης κρίσης που ζούμε σήμερα και με εξειδικευμένο τρόπο στο ανθρώπινο δυναμικό και γι' αυτό υποστηρίζουμε αυτή την πρόταση. Δεν υπάρχει επιστήμη χωρίς επιστήμονες και δυστυχώς έχουμε πολύ μεγάλες ανισότητες πολλές φορές. Μια άλλη παρατήρηση όσον αφορά την συνέχεια για την έρευνα και όσον αφορά τις κοινωνικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες ε, τι πρέπει να γίνει. Πιστεύω ότι εδώ ένα από τα αίτια θα μπορούσε να μας κάνει να συμφωνούμε. Εγώ συμφωνώ με αυτή την ε, κατανομή, με, αυτή, με αυτόν τον διαχωρισμό και για την ε, έρευνα για την ασφάλεια, όχι μόνο υπό την τεχνολογική πτυχή, είναι σημαντικό. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε μια συνέχεια στην αλυσίδα της έρευνας, θα πρέπει εδώ να ξεχωρίσουμε αυτά τα θέματα που είναι ξεχωριστά και που είναι ιδιαίτερη σημασία για τις κοινωνίες μας. Και τα θέματα των ανθρωπιστικών επιστημών ανήκουν σε όλες αυτές τις προτεραιότητες που έχουμε εντοπίσει. Δεν θέλω να μακρηγορήσω στην παρέμβασή μου, θέλω μόνο δύο ή τρεις παρατηρήσεις να κάνω πολύ σύντομα για θέματα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτα απ' όλα για τη σημασία της κατανομής των υποδομών και είναι θεμελιώδους σημασία να λάβουμε υπόψη ότι για να έχουμε ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα στην κλίμακά του, πρέπει να έχουμε αυτή την ευρύτερη διάσταση των υποδομών σε όλες τις χώρες, σε όλα τα κράτη-μέλη, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Είναι προφανές, ε, δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματα εξάπαντος, αλλά πρέπει να υπάρξει μια προσέγγιση και να υπάρξει καλύτερο συντονισμός μεταξύ των τριών πυλώνων. Να μην έχουμε τρία προγράμματα μέσα στο ίδιο το τελικό πλαίσιο, ενώ θα μπορούσε να είναι μέσα στον ίδιο πυλώνα ή να εντάσσονται στον ίδιο πυλώνα. Η ενίσχυση τέλος της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμφωνώ σε γενικές γραμμές με αυτά που προτείνονται και για τα μέσα αν υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες ούτως ή άλλως και δεν θα μακρηγορήσω λοιπόν πάνω σε αυτή την πτυχή. Προφανώς υποστηρίζω την διατήρηση των πόρων, αλλά με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και περνάμε τώρα σε εκείνους που πρόσεξε ο Πρόεδρος ότι ήθελα να παρέμβουν. Και η κυρία Γκροστέτ προστίθεται. Δεν είναι βέβαια κυρίες πρώτα, αλλά αυτή είναι η σειρά με την οποία σημείωσα. Ο κύριος Βίνταρ Κουάντρας, πρώτος δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι αυτονόητο ότι τα πρώτα μου λόγια πρέπει να είναι για να συγχαρώ τους εισηγητές και εισηγήτριες για το έργο που επετέλεσαν. Το πρόγραμμα για τον χρονορίζοντα 2020 με την ίδια την περιπλοκότητα των εγχειρημάτων και πρωτοβουλειών που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να καλύπτουν πολλές διαφορετικές πτυχές με ένα ενιαίο πλαίσιο επικέντρωσης και εστίασης όσον αφορά τις προτάσεις. Γι' αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο φαντάζομαι να αντιμετωπιστεί όλη αυτή η μάζα πληροφοριών και να εναρμονίσουμε τα πολλά διαφορετικά συμφέροντα μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα να επικεντρώσω τα σχόλιά μου για την πολύ καλή έκθεση που συνέταξε η κυρία Ριέρα Μαντουρέλ και που συμπεριλαμβάνει πολλές ε, πτυχές που αναφέρθηκαν στις συζητήσεις για τη δέσμη μέτρων για τον ορίζοντα 2020. Πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή έρευνα και η επισήμανση ότι τουλάχιστον το 15% των συνολικών προϋπολογισμών πρέπει να στοχεύουν ακριβώς σε αυτόν τον στόχο και για την υπενθύμηση ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής 2020 είναι αναγκαίο να προσφέρουμε κίνητρα στους ε, ε, ερευνητές στην Ευρώπη ώστε τα ταλέντα να μπορέσουν να προσελκυστούν και να έρθουν να συνεργαστούν, να εργαστούν στην Ευρώπη μαζί μας και για την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενημερώνει, να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το πρόγραμμα και υπάρχει η ανάγκη να υπάρχουν συμπληρωματικές δράσεις, παραπληρωματικές δράσεις και συνέργειες για την πολιτική συνοχή και για τον σημαντικό ρόλο των τοπικών αρχών και περιφερειών και περιφερειακών αρχών για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς πρέπει να αποφύγουμε την ε, περίπλοκη δομή των ε, γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων. Στην έκθεση της κυρίας Καρβάλιο έχουμε πάλι κάποια στοιχεία που πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι σημαντικά. Και με την διαφορετική εστίαση η αναζήτηση ενός καλύτερου συντονισμού για τον ορίζοντα 2020 και των διαθεωτικών ταμείων και τις δράσεις τους τίθεται το βάρος στη συμμετοχή της ευρωπαϊκής, ε, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην έρευνα καθώς επίσης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η προαγωγή, η προώθηση για να υπάρξει αυτός ο χώρος, ευρωπαϊκός χώρος έρευνας. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Well done. Thank you very much. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τσουκαλάς επόμενος. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτενείς ευχαριστίες στις εισηγήτριες σύντομα σχόλια επί του αντικειμένου. Άκουσα την κυρία Μαντουρέλ και θα συμφωνήσω μαζί της είναι απαραίτητη η άνετη χρηματοδότηση του προγράμματος. Αρχίσαμε από 100 δισεκατομμύρια, πάμε στα 80 δισεκατομμύρια, καταλαβαίνω ότι και εκεί θα υπάρξουν δυσκολίες δεν μπορεί να έχουμε μια κεντρική πολιτική και η κεντρική πολιτική είναι έρευνα και καινοτομία και ταυτοχρόνως να μην μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε με επάρκεια την κεντρική φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να θυμίσω ότι κατά τη δική μου αντίληψη η υποχρηματοδότηση της έρευνας δεν αποτελεί, δεν είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσεως η οικονομική κρίση είναι αποτέλεσμα του ότι δεν πετύχαμε το στόχο του 3% της στρατηγικής της Λισαβόνας. Φανταστείτε αν το είχαμε πετύχει τι θα γινόταν. Τώρα το αναβάλουμε μέχρι το 2020. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί πάνω σε αυτό. Φαίνεται ότι εάν η Ευρώπη συγκριθεί σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την καινοτομία και την τεχνολογία, δεν φαίνεται να κερδίζει αδάφος αλλά μάλλον να χάνει. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, καθώς επίσης πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι τα διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία μάλλον χρησιμοποιούνται κατά παράδοξο τρόπο στα διάφορα κράτη-μέλη, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά συζευκτικό τόπο, τρόπο με την γενική αντίληψη του ορίζοντα 2020 για να μπορέσουν να παραγάγουν αυτό που εγώ αποκαλώ όχι μόνο ε, R&D production αλλά R&D consumption as well. Τέλος, σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνητικών προσπαθειών ε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σκεφτεί την open access ως το αυτονόητο δικαίωμα του Ευρωπαίου πολίτη να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα έρευνας που χρηματοδοτήθηκαν από τα λεφτά του. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που σας βιάζω, συνάδελφοι. Ξέρω ότι σας απογοητεύει όλους, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Κύριε Αντελκαστήγιο, κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα, ξέρω ότι μίλησα ξανά, αλλά μίλησα εξ ονόματος του Κρίστιαν Έλλερ. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα. Καταρχάς, να συγχαρώ Εξ ονόματός μου τώρα, γιατί προηγουμένως ε, συνεχάρινε εκ μέρους του αδέλφου και, τους και τις εισηγήτριες και τους και που έκανε εξαιρετική δουλειά. Και θα σταθώ σε δύο θέματα απλά και συγκεκριμένα. Πρώτον, η διεθνή συνεργασία. Η κυρία Ρέιρα Μαντουρέλ το ανέφερε ως εγκάρσιο στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να ενταχθεί και στους τρεις πυλώνες του ορίζοντα 2020. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι προκειμένου να ενισχύσουμε ακριβώς αυτή τη στρατηγική, θα έπρεπε ίσως να υπάρξει ένας ορισμός ε, ενός ποσοστού δράσεων και κάποιων ελάχιστων στόχων, ώστε να μην είναι έτσι λόγο αλλά να είναι πιο συγκεκριμένο. Και κατόπιν για τις υποδομές έρευνας, κατά την άποψή μου θα έπρεπε να υπάρχει ένας, μια δυνατότητα αναβάθμισης, βελτίωσης των επιστημονικών μέσων και των πανευρωπαϊκών υποδομών που είναι υπαρκτή αυτή τη στιγμή, ε, το οποίο θα ήταν πολύ δύσκολο να το συμπεριλάβουμε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Νομίζω ότι αυτό θα βελτιώσει την επιστημονική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων. Αυτές οι δύο προτάσεις λοιπόν από πλευράς μου και φαντάζομαι ότι θα υπάρχει χρόνος να συζητήσουμε κάποια άλλα πράγματα περαιτέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Προφανώς δεν ήσασταν, ε, ε, δεν μιλούσατε εκ μέρους του κυρίου Ρέιλερ. Κυρία Νίμπλερ τώρα έχει τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Και εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ξεκινώ ευχαριστώντας θερμά την εισηγητρία, την συνάδελφο κυρία Ριέρα Μαντουρέλ και την κυρία Καρβάλιο. Πραγματικά σημαντικά θέματα έθιξαν και υπογράμμισαν πώς θα πρέπει να ε, τονιστούν και να συζητηθούν αυτά τα πράγματα από πλευρά του Κοινοβουλίου. Είμαι καταρχήν υπέρ της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υποστηρίζω όσον αφορά την θεμελιώδη προσέγγιση που έχει, αλλά και για το πρόγραμμα έρευνας βρίσκω καλές τις προτάσεις δεν είμαι κάποια που, ένα ε, άτομο που επενεί καθημερινά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γι' αυτό θέλω να το τονίσω. Επενώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια καλή πρόταση. Τι εξή προτάσει θα ήθελα να θέσω και θα ήθελα να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Το ένα είναι η ενιαία προσέγγιση και υποστήριξη για τι ε, βιομηχανίε, τι επιχειρήσει, μικρομεσαίε επιχειρήσει. Μέχρι στιγμή είχε ρυθμιστεί διαφορετικά το θέμα και θέλω να ρωτήσω, έχει νόημα πραγματικά κλιμακούμενα εδώ άσχετα σε ποιο θεσμικό όργανο αυτό εντάσσεται ή υπάγεται στην πρακτική εφαρμογή οδηγεί αυτό βέβαια ακριβώς οι βιομηχανικοί κύκλοι να την χάνουν επιπρόσθετα, επιπρόσθετων κονδυλίων για την έρευνα, ενώ ερευνητικοί φορείς υφίστανται περιορίσεις ή φοβούνται περικοπές και περιορισμούς. Και από τις συζητήσεις με τη βιομηχανία βλέπω ότι κατά πρώτη γραμμή δεν πρόκειται μόνο για τα κονδύλια για την έρευνα, αλλά και για το Ευρωπαϊκό Διεθνές Δίκτυο, που με την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα υποστήριξης μπορεί να προαχθεί. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω ποιες είναι οι απόψεις των συναδέφων για αυτά τα θέματα. Έχω επιφυλάξεις, αν μήπως δεν θα έπρεπε να παραμείνουμε στο πλαίσιο όσο είχε μέχρι σήμερα ποσόστοση και τρόπος υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 15% καταρχήν ερώτηση δεν θα μπορούσε να αυξηθεί αυτό το ποσοστό ενδυνάμωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πιέζει ο χρόνος θέλω να μιλήσω για το θέμα του πολιτισμού και της πολιτισμικής κληρονομιάς και την έρευνα για αυτό το θέμα. Δεν έχει ενταχθεί και θα ήθελα με τροπολογίες να το επανεντάξουμε. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ κυρία Γκροστέτ. Έχετε τον λόγο. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη για την έκθεση της κυρίας Μαντιουρέλ. Εκεί βλέπουμε πολύ θετικά πράγματα, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσουμε κυρίως το θέμα της αριστείας, που είναι απαραίτητο στοιχείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημιουργία πόλων αριστείας θα πρέπει να στηριχτεί οπωσδήποτε. Βεβαίως υπάρχει βούληση απλούστευσης των πραγμάτων έτσι ώστε ε, η δέσμευση και η συμμετοχή να είναι μεγαλύτερη. Γι' αυτό είναι καλό, αλλά βεβαίως θα πρέπει να το πετύχουμε. Θα ήθελα απλώς να εκφράσω την λύπη μου. Οι διεθνείς συνεργασίες, συνεργασίες δεν αναφέρονται πολύ στην έκθεση κυρίας Μαντουρέλ και λυπούμε γι' αυτό γιατί φρονώ είναι σημαντικό ε, να αφορούν αυτές οι συνεργασίες ε, προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κυρίως όταν μιλάμε για την έρευνα για μολυσματικές ασθένειες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για την έκθεση κυρίας Καρβάγιο, και εδώ έχω κάτι που με δυσαρεστεί, δηλαδή θεωρώ ότι η αναφορά στον τομέα της υγείας δεν είναι πάρα πολύ σημαντική ε, στην ε, έκθεση αυτή. Υπάρχουν βέβαια τροπολογίες οι οποίες προσπαθούν να αποζημιώσουν ε, αυτή την έλλειψη. Επίσης σημαντικό είναι να διατηρηθεί η χρηματοδότηση αυτό το 3% του ε, ΑΕΠ σε ε, ε, έρευνα και ανάπτυξη αυτή τη στιγμή γιατί έχουμε μπει πλέον σε φάση υπό επένδυσης. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά ο κύριος Ρογιάννα. Κύριε Πρόεδρε, είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα υπό την δική σας Προεδρία να μπορώ να παρέμβω με αυτή την παρέμβασή μου. Για το θέμα της έρευνας θα ήθελα να κάνω την εξή επισήμαση. Αν αληθεύει ότι έχουμε περιορισμένα κονδύλια και θέλουμε να πετύχουμε μέγιστο αποτέλεσμα και ταυτόχρονα έχουμε τη φιλοδοξία να προαγάγουμε την βέλτιστη έρευνα και να μην έχουμε την μέθοδο ε, δια του ε, με τα περιορισμένα κονδύλια να δρούμε. Τι θα κάνουμε για εκείνες τις περιοχές όπου η αριστεία δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα. Προσπάθησα σε σχέση με τις διαβουλεύσεις, να προσελκύσω και να βρούμε ένα τρόπο να διαθέσουμε κονδύλια για τον ανταγωνισμό. Ανταγωνισμό και συναγωνισμό όπου μια βέλτιστη ε, αριστείας προσέγγιση θα συνδέεται με ένα θεσμικό όργανο για ένα πεδίο που μέχρι σήμερα δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα επιστημονικά. Και αυτός ο ανταγωνισμός ή συναγωνισμός να αξιολογείται και να υπάρχει υποστήριξη μετά για τις βέλτιστες προσεγγίσεις. Αυτό θα μπορέσει να δώσει την δυνατότητα να έχουμε, πράγμα το οποίο εξέθεσε συνάδελφος, και την χρήση των διαθροτικών ταμείων, των κονδυλίων των διαθροτικών ταμείων και των κονδυλίων για την έρευνα. Δηλαδή αριστεία για τους τομείς εκείνους που πρέπει να προαχθούν ιδιαίτερα. Και θα είμαστε πιο δίκαιοι για τα θέματα που έθιξαν συνάδελφοι από τα κράτη-μέλη που δεν διαθέτουν και δεν την χάνουν πολλών κονδυλίων για αυτές τις δράσεις. Και έτσι θα μπορούμε να προαγάγουμε μόνο εκείνα τα οποία ανταποκρίνονται στην αριστεία και δεν θα δίνουμε ισοπεδωτικά κονδύλια σε όλους ε, ε, που είναι και περιορισμένα. Έτσι θα μπορέσουμε με καλύτερο στοχοθετημένο τρόπο να διαθέσουμε τα περιορισμένα μας κονδύλια. Διότι υπάρχει το αίτημα αυτές τις ημέρες να, να ανταποκριθούμε στο εύρος των αναγκών της Ευρώπης και να μην μείνουμε πίσω. Ευχαριστώ. Um, Mr. Skinner, you said you only... Σας ευχαριστώ. κύριο Σκίνερ τώρα. Um, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τις εισηγήτριες. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια που ακούστηκαν όμως μερικά ε, όσον αφορά την κλίμακα αριστείας ε, δεν μπορούμε ε, να ξεχωρίσουμε αυτή την κλίμακα αριστείας και από το θέμα της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας. Ξέρουμε ότι επίσης η βασική έρευνα τι σημαίνει βασική έρευνα. Οι μόνες θέσεις που εργασίας που μπορούν να δημιουργηθούν είναι μονάχα στα εργαστήρια. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε εάν αποφασίσουμε τελικά να οθήσουμε μόνο την βασική ε, έρευνα. Ε, οι κλίμακες αριστείας είναι αυτές οι οποίες προσεγγίζουν την αριστεία της ε, αγοράς και θα πρέπει να τις στηρίξουμε. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που οι συγγήτρες είναι αυτές που είναι. Ξέρω ότι και η κυρία Μαντουρέλη και η κυρία Καρβάγιο θα βοηθήσουν έτσι ώστε τα πράγματα να προχωρήσουν καλά. Εξαιρετικά. Λοιπόν, ο κύριος Μπούζεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής ε, γιατί έχουμε αυτήν την συζήτηση με τόσες ενδιαφέρουσες προτάσεις για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο και για τον ορίζοντα 2020. Συγχαρητήρια για τις εισηγήτριές μας ε, και τις δύο. Είναι πάρα πολύ καλή η δουλειά σας. Κάνατε εξαιρετικές εκθέσεις. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω των εκπροσώπων τους εδώ. Γιατί ένα από τα πιο δύσκολα σημεία, θέματα, 7 ε, χρόνια πριν, ε, ήταν ακριβώς ε, η διάχυση και η διάδοση της αριστείας και η ενίσχυση της συμμετοχής, δηλαδή μεγαλύτερη συμμετοχή χωρίς όμως να πέσει το επίπεδο της αριστείας. Είχαμε αρκετή επιτυχία στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και τώρα αναφέρονται και κάποιες συγκεκριμένε προτάσεις. Ε, επομένως, ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς το Συμβούλιο. Ε, τέσσερις είναι οι προτάσεις. Πρώτον, στην συνέργεια μεταξύ των διαθετικών ταμείων και των ε, του ορίζοντα 2020, ε, γνώση της ε, συμμετοχής. Δεύτερον, αν ελεύθερη ανοιχτή πρόσβαση και ετικέτα αριστείας. Τρία, μικρομεσαία προγράμματα αυτό βεβαίω εμπλέκει τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Είναι ένα άλλο τρόπο για να αναφερθεί κανεί στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Πώ μπορεί, μπορεί κανεί να στηρίξει και να προωθήσει τέτοια πράγματα. Και τελευταίο, τέταρτο τελευταίο σημείο. θα πρέπει να βρεθεί μία φόρμουλα για το, α, για το κόστος ε, ανα ε, μονάδα, έτσι ώστε να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Η ίδια προσέγγιση η οποία, ε, την οποία είχαμε εις, το, θέμα της κινητικότητας. αν μπορούσε κάποιος να απαντήσει σε ερωτήσεις μου θα ήταν πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπούζεκ, ο Πρόεδρος. Είσαστε όλοι πάρα πολύ καλοί μαθητές. και επομένως ε, έχει περισσέψει λίγος χρόνος και επομένως μπορώ να δώσω, εάν θέλουν οι εισηγήτριες, λίγο χρόνο. Ε, κυρία Καρβάγιο, αν θέλετε πρώτα στην κυρία Μαντουρέλ. Ναι, απευθύνθηκα πρώτα στην κυρία Καρβάγιο, γιατί εσείς μιλήσατε περισσότερο χρόνο στην αρχή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, χαίρομαι που έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Θα ήθελα να απαντήσω λίγο σε όλους όσους ε, έλαβαν το λόγο και να σας ευχαριστήσω όλες και όλους ε, για τη συνεισφορά σας, για τον ενθουσιασμό σας και για το ενδιαφέρον σας, ε, διότι σημείωσα πολύ καλά όλα όσα άκουσα. Ε, πολλά πράγματα βέβαια τα είχαμε συζητήσει και απευθείας και είναι βέβαιο ότι σίγουρα θα τα και στην τελική μου έκθεση. Αναφέρθηκα προηγουμένως στην εξαίρετη συνεργασία με τους κοιόδης συζητητές και με ε, τη, επειδή συζητήσαμε από κοινού και με την κυρία Καρβάγιο και τις δύο εκθέσεις, ε, θα ήθελα να επισημάνω πόσο καλή συνεργασία και καλό συντονισμό είχαμε με την κυρία Καρβάγιο. Η κυρία Καστίγιο που μίλασε εξ του κυρίου Έλερ είπε αρκετά πράγματα τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να τα συζητήσω και με τον κύριο Ελέρ, αλλά επισήμανε για άλλη μια φορά και πόσο σημαντικό είναι ο προπολογισμό. Να υπάρχουν αρκετά χρήματα για να τεθεί σε εφαρμογή το ορίζον 2020. Αυτό είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, αν πραγματικά θέλουμε να εφαρμόσουμε τη στρατηγική του 2020. Δεν θέλω να επισέλθω σε περισσότερε λεπτομέρειε, αλλά νομίζω ότι το συνειδητοποιούμε όλοι πώ έχει το ζήτημα. Όσον αφορά την ισότητα των φύλων, ε, το οποίο ε, θέσατε επίση, είναι ένα από τα σημεία τα οποία δεν μπορεί να σχολιάσω στην αρχική μου παρέμβαση, διότι μία από τις πτυχές και ένας από τους λόγους που μας ε, παρακίνησαν ήταν ακριβώς ε, και το γεγονός ότι θα θέλαμε να επισημάνουμε τον παραδειγματικό χαρακτήρα του προγράμματος και γι' αυτό ακριβώς ε, θέλαμε να καταθέσουμε και τροπολογίες για την ισότητα των φύλων. Θεωρούμε ότι το ορίζον 2020 θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα και Ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει κατά την άποψή μου και ένα άρθρο το οποίο θα είναι αφιερωμένο στην ισότητα των φόλων. Και με τις τροπολογίες μου έχω αναφέρει τη διπλή πτυχή του ζητήματος. Καταρχάς να αυξηθεί η αντιπροσώπευση των γυναικών ε, στη στρατηγική και στην Ευρώπη 2020, αλλά ταυτόχρονα να δώσουμε και νέα έφεση στην έρευνα και τις μελέτες για θέματα φύλων. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στο γεγονός ότι έχουμε συμπεριλάβει και ένα νέο άρθρο το οποίο μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε ε, κάποιο σχόλιο που ακούστηκε και κάποιον, από κάποιον άλλον από τους ομιλητές ε, την ανοιχτή πρόσβαση στις δημοσιεύτες και στα αποτελέσματα της ε, έρευνας η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 και τη δυνατότητα να προωθήσουμε αυτή την ανοιχτή πρόσβαση στα στοιχεία τα οποία λαμβάνονται από προγράμματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το Horizon 2020. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να απαντήσω σε όλους, αλλά βλέπω ότι δεν θα μου δώσετε τόσο χρόνο. Να σας πω λοιπόν απλώς ότι σημείωσα όλα όσα είπατε και αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία θα το συζητήσω διαζώσεις ε, μεταξύ ε, μας και σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοι θα χαρούν με την προσφορά σας να συζητήσετε τα θέματα διμερώς. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Καλβάγιο, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα δώσουμε το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος ε, του τρίτου τμήματος αυτής της κοινή συζήτηση. Αν νομίζετε λοιπόν ότι τους έχω παραβλέψει, δεν τους έχω παραβλέψει. Θα ε, ακούσουμε την Κομισιόν στο τέλος, θα μας τα πει όλα. Κυρία Καλβάγιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου για τα σχόλια που έκαναν. Βεβαίω δεν θα απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά. Θα ήθελα απλώ να υπογραμμίσω κάποια από τα σημεία. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην διεύρυνση της συμμετοχής. Είναι ένα θέμα το οποίο ιδιαίτερος πρόσεξα στην έκθεση και οι προτάσεις ε, που υπέβαλε και οι ερωτήσεις που υπέβαλε ο πρόεδρος Μπούζεκ στην ε, Κομισιόν αναφέρονται ήδη στην εκθεσή μου, δηλαδή καλύτερη συμμετοχή, καλύτερη ισορροπία μάλλον όσον αφορά τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η πρόσβασή τους Ε, τώρα όσον αφορά την, τις προτάσεις που ακούστηκαν, βεβαίως μπορούμε στη δεύτερη φάση των τροπολογιών να τις εντάξουμε. Διεθνή συνεργασία ε, βεβαίως ε, δεν αναφέρεται η διεθνή συνεργασία ιδιαίτερα ε, στην έκθεση κύρια Μαδουρέλα, αλλά στη δικιά μου ε, δίνονται και συγκεκριμένα παραδείγματα με στοχευμένες συνεργασίες για συγκεκριμένους τομείς, ας πούμε ενέργεια για τη Βραζιλία. Ε, προγράμματα καταπολέμησης ένδυας ε, σε συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες, τεχνολογική συνεργασία με τις Ηνωμένες την Νότια Αφρική, την Αυστραλία κλπ. Επομένως υπογραμμίζεται ιδιαίτερος η διεθνή συνεργασία. Uh, uh, όσον αφορά την ε, υγεία, ναι, είναι γεγονό ότι ε, δεν υπάρχουν πολλέ τροπολογίε όσον αφορά ε, την υγεία. Όμω, εγώ αναφέρθηκα ιδιαίτερα στην παρουσία των Ευρωπαίων ερευνητών σε τομεί υγεία και σε πολλέ τροπολογίε αναφέρεται ο τρόπο καλύτερου επιστημονικού συντονισμού της έρευνας για την υγεία στην Ευρώπη με τρόπον ώστε να μπορούμε να ανταλλάσσουμε ε, πληροφορίες, στοιχεία κλπ έτσι ώστε ε, οι ε, μελετητές οι οποίοι εργάζονται για ορφανές ασθένειες, σπάνιες ασθένειες να μπορούν να συνεργάζονται με άλλους ερευνητές στις χώρες μέλη. Επομένως, ναι, έχουμε υπογραμμίσει και το θέμα της υγείας και θα γίνει πολύ συγκεκριμένο, μάλλον θα βρει το συγκεκριμένο του αντίκτυπο σε συγκεκριμένες ε, δράσεις, αλλά βεβαίως μπορούν να υπάρξουν περαιτέρω τροπολογίες ε, και γι' αυτό και για άλλα θέματα θα σας στείλω και όλα τα σχόλια. Uh, um, Ευχαριστώ πολύ και ολοκληρώσαμε λοιπόν την συζήτηση για την πρώτη ομάδα εκθέσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, τις εισηγήτρες ιδιαιτέρως, αλλά και όλους όσους πήραν το λόγο, χωρίς να ξεπεράσουν τον χρόνο τους. Λοιπόν, θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, κυρία Ματράς. Do minutes. Ε, στην κυρία Ματία, συγγνώμη. Ε, παρακαλώ να μην ξεπεράσετε το χρόνο σας. Έχετε το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα και εγώ επίσης θέλω να πω θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία όλων των συνάδελφων στην εκπόνηση αυτής της πρώτης πρότασης μετά τις ανταλλαγές που είχαμε απόψεων καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου και θέλω να πω ότι πρόκειται για μια πρόταση που προφανώς από την πρόταση του κυρίου Λαμπέρτ συνεξετάστηκε και ως μέρος ε, και της ατζέντα του θεματολογίου της ε, καινοτομίας ε, για την έρευνα. Θέλω να επικεντρωθώ σε αυτά που είναι οι κυριότερες προτάσεις αυτού του θεματολόγιου για την καινοτομία όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Πρώτα για τον τύπο και μετά για την ουσία για την, τον τύπο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ένα άρθρο στο νομοθετικό σκέλος που θα πρέπει να εγκρίνει αυτό το οποίο εντάσσεται στο παράρτημα. Η δική μου εναλλακτική λύση ήταν, και το εξηγώ αυτό, να θέσω μια αιτιολογική σκέψη για τα κυριότερα στρατηγική σημασία θέματα στην αρχή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θεματολόγιο. Στην αρχή αρχή τέθηκε για να ξεχωρίσουμε τις προτεραιότητες ε, της παρέμβασης όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία και μετά μπορούν να υπάρξουν τροποποιήσεις στο παράρτημα σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, με αυτόν τον τύπο. Υπό γενικού όρου, τι προτείνεται σε αυτή την έκθεση. Μέχρι σήμερα είχαμε ένα ίδρυμα το οποίο λειτουργήσε κυρίως ως συγχώνευση τριών ενωτήτων για την ενέργεια, τις κλιματικές αλλαγές, για τις, ε, την επικοινωνία. Έχουμε μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που την υποστηρίζω να αυξηθεί ο προϋπολογισμός μας ε, όσον αφορά τα κονδύλια που διαθέτουμε και το εγκρίνω αυτό. Αυτή η αύξηση θα πρέπει να υποστηριχθεί. Χρειαζόμαστε πραγματικά αυτό το Ίδρυμα και όχι μόνο μια συνάθρηση των τριών κοινοτήτων ή τριών δράσεων. Ένα αυθεντικό Ίδρυμα, ένα Ινστιτούτο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να εξεταστούν και άλλα θέματα φυσικά. Αυτονόητο, αυτονόητο είναι ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας είναι το μόνο μέσο που μπορεί να αρθρώσει τη γνώση ε, και τις ε, ανάγκες που απορρέουν από τη γνώση από τα πανεπιστήμια μέχρι την έρευνα. Να είναι το μέσο το οποίο θα έχει τη μεγαλύτερη επιστροφή, τη μεγαλύτερη πρόσθετη αξία. Με τη χρηματοδότηση ε, δημόσια και ιδιωτική θα έχουμε πολύ μεγάλη επιστροφή και πρόσθετη αξία για τις μονάδες που θα ε, συμμετέχουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να υπάρχει μόχλευση δηλαδή, να υπάρξει μοχλική επίπτωση. Θα πρέπει να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε, κινητοποιήσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία με αυτή τη μόχλευση. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστούν λοιπόν αυτές οι πτυχές μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Επιπρόσθετα, οι κοινότητες γνώσης και οι κοινότητες, ε, ερευνητικές κοινότητες γνώσης θα πρέπει να επεκταθούν σε περαιτέρω συνιστώσεις που πρέπει να προσθεθούν. Φυσικά μια προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στην κατάρτιση και εκπαίδευση και εδώ υπάρχει και η δυνατότητα, η πρόταση να υπάρξει ένα πρόγραμμα υποτροφιών για την έρευνα. Υποτροφίες που θα δίνουμε για να διευρυνθεί η δυνατότητα για, τα, για τις ερευνητικές δραστηριότητες μέσω του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Και μια συγκεκριμένη πρόταση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Να υπάρχει δηλαδή συνάρτηση με την απασχόληση νέων επιστημόνων που ε, με προγράμματα που θα συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα τεχνολογίας να υπάρχει δυνατότητα για αυτούς τους επιστήμονες ένα μέρος, ένα τμήμα αυτών να μπορούν να απασχοληθούν, να μπορεί να δοθεί δραστηριότητα σε αυτούς όσον αφορά την απασχόληση. Αυτό είναι σημαντικό για αυτούς τους τομείς έρευνας. Από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ένας τομέας που πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα αυτός. Μία άλλη παρατήρηση για να πω ότι πρέπει να έχουμε, να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή. Έχουμε συγκεκριμένα εξειδικευμένα στρατηγικά μέτρα και πρωτοβουλίες ώστε οι μονάδες, οι οι δυνατότητες ε, διάδοσης και διάχυσης της γνώσης να μπορούν πανευρωπαϊκά να δράσουν. Και πρέπει να μπορούμε να κινητοποιήσουμε αυτές τις μονάδες και όχι να παραμένουμε σε, λίγα, σε κάποιες λίγες έδρες που θα ε, δρουν στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχέονται οι δυνατότητες συμμετοχής μέσω αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας. Τούτων λεχθέντων θα πρέπει να δούμε και κάτι το οποίο απουσίαζε, όχι μόνο επειδή δεν είχε ξεκινήσει, επειδή όμως λείπουν και κάποια στοιχεία για να μπορούν να, να, να δρουν όπως ε, το επιθυμούμε. Και πρέπει να έχουμε το πρόγραμμα αριστείας και βέλτιστης απόδοσης όσον αφορά την έρευνα. Και αυτά τα οποία αναφέρθηκαν για τον ορίζοντα 2020, τον χρονορίζοντα, χρειαζόμαστε διαφορετικές υποδομές. Θα πρέπει να δημιουργηθούν αυτές οι υποδομές σε αυτό το χρονορίζοντα. Και η πρόταση είναι να υπάρξει ένα άρθρο το οποίο θα ζητεί ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ίδρυμα να μελετήσουν τη δυνατότητα να, έχουν την έδρα, να έχει την έδρα του στο Στρασβούργο το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ίδρυμα. Και το επεξηγώ αυτό με ένα λόγο πολύ απλό. Σήμερα το Στρασβούργο είναι περισσότερο ένα πρόβλημα και όχι λύση για τους πολίτες μας ενώ με το οριζόντιο εγκάρσιο πρόγραμμα του ορίζοντα 2020 και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας θα υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει πρόσθετη αξία με ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα το οποίο θα δίνει αυτή την πρόσθετη αξία με έδρα το Στρασβούργο. Με αυτό και ακριβώς με εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε υπέρ του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Ιδρύματος πρέπει να μεταμορφώσουμε τη συμβολική αυτή, ας το πω, το τη συμβολική εικόνα από αρνητική σε θετική. Είναι θετικό λοιπόν το Στρασβούργο και μπορεί να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη θετική απήχηση αν θα είναι η πρωτεύουσα της καινοτομίας και της ε, γνώσης. Και με το κέντρο αριστεία στην Ευρώπη, με την έδρα που θα έχει στο Στρασβούργο το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας. Θα πρέπει να δούμε Πώς είναι δυνατόν να έχουμε κτίρια τα οποία μόνο τρεις ή τέσσερις ημέρες θα απασχολούμε και βρισκόμαστε σε αυτά ε, κάθε μήνα. Πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Υπό αυτό το πρίσμα υποβάλλεται αυτή η πρόταση. Για το μέλλον πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα που θα προβάλλουμε ως προοπτική. Ένα σύμβολο ευρωπαϊκό με έδρα το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ίδρυμα στο Στρασβούργο. Έτσι πρέπει να έχουμε το θάρρος να σκεφτούμε για το μέλλον με μια προοπτική τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για την Ευρώπη στο μέλλον, για την καινοτομία και τη γνώση. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν αντί να δίνουμε μάχες κατά του Στρασβούργου πρέπει να επενδύσουμε στο Στρασβούργο για την τεχνολογία και την αριστεία της έρευνας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας άφησα να ξεπεράσετε το χρόνο. Α, α, μόνο γιατί ίσως μου άρεσε η ιδέα ότι ίσως δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουμε στο Στρασβούργο πια. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Λαμπέρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη που έφτασα αργά, ήμουν στην ΕΚΟΝ. Ε, δεν ήταν ότι έπαιρε την πυρίτσα μου έξω. Λοιπόν, ε, για τα επόμενα 55 λεπτά μπορώ να εξηγήσω, για, να μιλήσω για έκτη φορά για την έκθεσή μου. Όχι, καλά. Λοιπόν, ε, ήδη γνωρίζουν όλοι και νομίζω και οι σκιώδεις ε, τις ιδέες μου. Θα ήθελα παρόλα αυτά να υπογραμμίσω κάποιες ιδέες που έχω για την ε, ε, συνολική δέσμη, για το πακέτο γιατί είμαι και εισηγητής και ταυτόχρονα σκιώδης για, όλο το, για όλη τη δέσμη. Ε, πρώτα απ' όλα, ε, εγώ δεν θέλω να ξεκινήσω μάχες ε, με τους ε, ε, και με τους συναδέλφους. Είμαι μάλλον άνθρωπος της σύνθεσης. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα πρώτο στοιχείο που έχω υπογραμμίσει, ε, το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Ε, θα ήθελα περισσότερη ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και λέω ότι αντί να επιλεγούν κάποια στοιχεία όπως κάνει η Κομισιόν να βάλουμε δίπλα-δίπλα τα στοιχεία και το καλύτερο ας κερδίσει. Δεύτερον, ε, μιλήσαμε για αμόχλευση. Ε, είπαμε ό μάλιστα το αναφέραμε και στην ε, προηγούμενη συνεδρίαση των σκιωδών. Ξέρετε ότι αυτός ο κανόνας του 25% υπάρχει. Εμείς θα θέλαμε σε ολόκληρο το πρόγραμμα να υπάρχει μια τέτοια αντιμετώπιση ε, θα ήθελα λοιπόν να δω από μη ευρωπαϊκές πηγές να έρχονται χρήματα ε, προς, αυτό το πρόγραμμα. Γιατί εάν το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά με ευρωπαϊκά χρήματα, τότε ίσως, ίσως θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν είναι πραγματικά ένα καλό πρόγραμμα. Κατά αυτή την έννοια θα ήθελα ένα ε, ε, ευρώ, ε, ένα ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσθεθεί σε πολλά ευρώ από άλλες πηγές. Θέλουμε επίσης άλλο σημείο, θέλουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όχι μονάχα για τη μόστρα, για τη βιτρίνα. Θέλουμε πραγματική συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το 15% στο 20% και παραπάνω. και όσοι στον ιδιωτικό τομέα έχει δουλέψει και με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με μεγάλες πολυεθνικές ξέρει ότι δεν μιλάς με την IBM με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο μιλάς ε, με τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή θα πρέπει να ε, ξέρει κανείς με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ποια γλώσσα θα χρησιμοποιήσει. Αυτά θα πρέπει να ισορροπηθούν, να υπάρχει μια ισορροπία και σε αυτά τα στοιχεία. Επίσης, θα θέλαμε να δούμε περισσότερα ε, στις κοινωνικές επιστήμες, ανθρωπιστικές σπουδές. Ξέρουμε ότι υπάρχει... Ε, εδώ, κοιτάξτε, ε, εδώ δεν είναι να δώσουμε έτσι ένα κομματάκι στις κοινωνικές επιστήμες και στις ανθρωπιστικές σπουδές έτσι ώστε να είναι ικανοποιημένες. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε ένα πραγματικό χώρο για αυτές τις σπουδές γιατί η τεχνολογία από μόνη η επιστήμη από μόνη μόνη της δεν μπορεί να δώσει ε, τις απαντήσεις ε, για όλα. Ε, γιατί βεβαίως θέλεις τεχνολογία έτσι ώστε να ανακυκλώσεις τα σκουπίδια σου, αλλά θέλεις και κοινωνικές αλλαγές και κοινωνική ευαισθητοποίηση έτσι ώστε να έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Επομένως θέλουμε ανθρωπιστικά κοινωνικά στοιχεία που θα προκύψουν από αυτές τις επιστήμες και από αυτή την έρευνα θέλουμε ανοιχτή κοινωνία ε, με ελεύθερη ροή της γνώσης. Θα πρέπει να δουλέψουμε καλύτερα όσον αφορά την διάχυση των αποτελεσμάτων ε, και όσον αφορά ε, την διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων. Γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε πραγματική πρόοδο και πραγματική καινοτομία. Εάν κανείς κρατήσει τη γνώση για τον εαυτό του, τότε δεν πρόκειται να επιτευχθεί τίποτα. Δεν λέω ελεύθερη γνώση για όλους. Λέω ότι θα πρέπει να ε, ενθαρρύνουμε την ελεύθερη ροή της γνώσης στην κοινωνία, έτσι ώστε να φτάσουμε πιο γρήγορα στην καινοτομία. Ε, θα μπορούσα να προσθέσω και κάτι για αυτήν την έκτη πρόσκληση ε, που παντρεύει την ασφαλή κοινωνία με την ανοιχτή κοινωνία. Ξέρω ότι μεταξύ ημών υπάρχουν αυτοί που θέλουν κάτι περισσότερο όσον αφορά την ασφάλεια, την γενοτομία και την ε, ε, ε άμυνα. Κοιτάξτε, δεν ξέρω γιατί δεν θα πρέπει να είναι δυνατή ε, η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Όχι, όμως νομίζω ότι θα πρέπει η άμυνα πρώτα να γίνει κοινοτική ε, αρμοδιότητα. Ε, μέχρι τότε όμως παραμένει μη κοινοτική, εθνική αρμοδιότητα. Άρα θα πρέπει να χρηματοδοτείται από, την εθνική, ε, από τις εθνικές αρχές και από την από τον εθνικό προϋπολογισμό. Έχουμε ήδη λίγα χρήματα, έχουμε 80 δις. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε να λύνουμε εθνικά θέματα χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκά χρήματα. Εάν ε, θέλουν κάποιοι να ε, βοηθήσουν ε, τους, την Εθνική του Μηχανία Άμυνας ή κάτι τέτοιο και την έρευνα, κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος και χώρος για αυτά τα πράγματα. Αυτά μίλησα για την έκθεσή μου τελικά μόνο και νομίζω ότι δεν ξεπέρασα το χρόνο. Με ευχαριστώ πολύ. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στους υπόλοιπους κοιόδης εισηγητές, ε, διότι θα δώσουμε το λόγο όχι μόνο στους εισηγητές, αλλά και στους κοιόδης. Ο κύριος Τσουκαλάς καταρχάς, σας δώσει το λόγο αν τον επιθυμείτε. Two minutes. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, λίγα πράγματα θα πω σχετικά με τις εκθέσεις για το EIT. Αντιμετώπισα μαζί με τον κύριο Βανίστερ Λόι τα οχτώ θέματα που αναφέρονται σε αυτές. Το πρώτο είναι ο προϋπολογισμός, το δεύτερο είναι οι κανόνες, το τρίτο είναι η έδρα, το τέταρτο είναι η επιλογή των ΚΙΚΣ, το έκτο είναι η χρηματοδότηση των ΚΙΚΣ, το έβδομο είναι η παρακολούθηση των ΚΙΚΣ, το όγδο είναι η συμπερίληψη των κοινωνικών επιχειρήσεων και του IPR και τέλος είναι το ένατο η διοίκηση των ΚΙΚΣ. Επί αυτών έχει διανεμηθεί το κατάλληλο κείμενο. Θέλω να σας πω ότι η άποψη μου είναι ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Η άποψη μου είναι ότι δεν πρέπει να περικοπεί ο προϋπολογισμός των ΚΙΚΣ όπως προτείνεται από την έκθεση της κυρίας Μαντουρέλ από το 3,64% στο 3,1% Επίσης νομίζω ότι η επιλογή των ΚΙΚΣ θα μπορούσε να γίνει με τον τρόπο που λέει ο κύριος Λάμπερτς με μικρές τροποποιήσεις. Δεν θα έπρεπε να δίνουμε χρήματα για τα ΚΙΚΣ εκεί και ως έλαχεν. Θα περίμενα μέχρι το, τα έξι καινούργια ΚΙΚΣ να γίνουν σε δύο κύματα 3 και 3 αφού προηγουμένως ελέγξουμε ποια είναι τα παραδοτέα με πολύ αυστηρούς ε, κανόνες. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε ε, μια ε, μέση λύση έτσι ώστε οι τροπολογίες που θα κατατεθούν να βοηθήσουν την βελτίωση των δύο εκθέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που τηρήσατε και τον χρόνο που σας διέθεσα. Ο κύριος Γιωχάνσεν στη συνέχεια, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την καλή συνεργασία και ελπίζω να υπάρχει και αποφωνία 90%. Και επίσης να πω Horizon. Όταν ε, πρωτοπροτάθηκε το Horizon 2020, ήμουν από τους πρώτους που πρότειναν αύξηση ε, του προϋπολογισμού για το EIT, αλλά, το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ίδρυμα, αλλά στη συνέχεια, βλέποντας τα διάφορα ερευνητικά κέντρα και συζητώντας και με τον κλάδο και τα ερευνητικά Ινστιτούτα, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ έρευνας και αγοράς. Ε, το λέει και κάποιος από τους συζητητές. Χαίρομαι λοιπόν για τον προπολογισμό για το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ίδρυμα και ελπίζω να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε κιόλα. Επίσης, ε, έθεσα και μία ερώτηση για τα διάφορα kicks και τη διαδικασία επιλογής των. Νομίζω ότι συμφωνώ ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτό και στα έξι θέματα τα οποία είχαμε ήδη μέχρι το 2014, διότι είναι πιο λογικό να βασίσουμε τις συζητήσεις επί του προπολογισμού για κάθε κικ ξεχωριστά και ε, όσα ε, μας δίνει και να μην τα συγκρίνουμε με την απόδοση ε, των υπολείπων κικς. Ε, ο ανταγωνισμό λοιπόν μεταξύ των από εκεί και πέρα θα είναι σημαντικό στοιχείο και από εκεί και πέρα θα δούμε και τι δυνατότητε του Τεχνολογικού Ιδρύματος και θα δούμε και πώς μπορούμε να τα προχωρήσουμε. Επίσης θα ήθελα να σχολιάσω και κάτι για τα θέματα ε, πνευματικών δικαιωμάτων και την ανοιχτή πρόσβαση. Νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει ένα από τα ε, πιο διαφιλονικούμενα ζητήματα προς συζήτηση Καλό είναι να γίνει συζήτηση. Εγώ θέλω να προασπίζονται τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά καλό θα ήταν να δούμε και τι γίνεται με τα ανοιχτή πρόσβαση και τις διάφορες πλατφόρμες που προσφέρουν ανοιχτή πρόσβαση. Ε, για την έκθεση της κυρίας Ματίας ε, τώρα, θα ήθελα να υπάρχει και μια διευρυμένη αποστολή της, ε, και για τα ΚΙΚΣ, ιδίω από την εκπαιδευτική τους πλευρά και με ανησυχεί λίγο το γεγονός αυτό, διότι ο προπολογισμό δεν ανταποκρίνεται σε αυτή τη διευρυμένη αποστολή. Θα μπορούσε να μας σχολιάσει λίγο το θέμα αυτό στη διάρκεια της συζήτησης ε, και να το διευκρινίσουμε στη συνέχεια μέσω τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Φανίστελ Ρόι τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Κάποιες ε, παρατηρήσεις Ευχαριστώ τις εισηγήτρες και του εισηγητές. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι τόσο πεισμένο για το Στρασβούργο. Τι στοχεύετε να πετύχετε. Νομίζετε ότι θα περάσουν σε μια άλλη κατεύθυνση κάνοντας το όχι ναι στη Γαλλία για τους Γάλλους με την τοποθέτηση αυτού του Ινστιτούτου εκεί. Και πώς είναι δυνατόν να ξεκινήσουν όλα αυτά. Είναι μια καλή έκθεση αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω πώς στοχεύεται σε κάτι τέτοιο. δεύτερο. πώς θα επιλεγούν τα kicks. Νομίζω θα πρέπει να μην χάνουμε χρόνο. Θα πρέπει να έχουμε μια ανοιχτή προσέγγιση ιστερότερα. Πρώτα στοχοθετημένα και μετά σε ένα πιο ανοιχτό πλαίσιο. Σε σχέση με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν στη συζήτηση για τη συμμετοχή από όλες τις πλευρές της Ευρώπης σε αυτό το πλαίσιο Χρειαζόμαστε κάτι πρόσθετο, κάτι ακόμα. Έχουμε τα κίξ και είναι κάτι αναγκαίο που πρέπει να υπάρχει εδώ, ώστε να προσφέρουμε το πολύ μεγαλύτερο δυναμικό και να αντλούμε από αυτό σε σχέση με τις ε, βιομηχανίες επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια. Αν δείτε μόνο την ακμή, την ε, ε, ακμή του τριγώνου δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις διαφορετικές δυνατότητες. Το να υπάρξει μια νέα δυνατότητα που θα μπορέσουμε να την ε, εκμεταλλευτούμε συνδέοντάς την ε, με άλλες ε, υφιστάμενες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλες υπαναχωρήσεις όσον αφορά την αριστεία και την υπέροχη. Να χρησιμοποιούμε περισσότερο εκείνα τα οποία είναι δεδομένα για παράδειγμα, σε σχέση με εκείνα τα οποία συμμετέχουν είτε πλήρως ή όχι στα ΚΙΚΣ και να δημιουργηθεί η δυνατότητα να υπάρχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα στο μέλλον. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Κύριε Λάμπερ, θέλετε ξανά το λόγο ως σκιώδης, όχι. Επομένως, να δώσω το λόγο τώρα ε, στον Σάντο από το ECR ή να δώσω το λόγο στον εαυτό μου ενδεχομένως. Να πω πολύ σύντομα, χωρίς να χαλάσω λίγο την ωραία ατμόσφαιρα, ε, να πω λοιπόν ότι δεν είμαι απολύτως πεπισμένο ε, για το επίτευγμα αυτό του EIT, του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Ινστιτούτου, θα πρέπει, Ιδρύματος, θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι καλό. Έχουμε δύο... Είμαστε νομίζω πολύ φιλόδοξη με τον προπολογισμό και πολύ φιλόδοξη με τα κίξη. Γι' αυτό λοιπόν θα, ε, βάλω, θα υποβάλω και κάποιες ε, τροπολογίες. Αυτά θέλω να πω, δεν έχω τίποτα άλλο, κύριε Καρβάλιο. Thank you very much. I would like to... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές ε, και, την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε όχι με όλους τους αδέλφους, όχι μόνο με τους σκιώδεις. Να τονίσω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε μία ε, ενιαία γραμμή ε, και με το θέμα του ορίζοντα 2020 και όσον αφορά και τη συνέργεια με, τους, ε, με τα διορθωτικά ταμεία, ε, με τα κέντρα αριστείας έτσι ώστε ε, να μπορούν να εφαρμοστούν ε, και στα IT όλα αυτά που αναφέραμε και πριν για τον ορίζοντα 2020 και για το IT. Δεύτερον, να υπογραμμίσω την ε, σημασία του EIT ε για την δημιουργία ε, βιώσιμων startups. Βεβαίως μπορούμε να το δούμε και για τα εκείξια, αλλά και σε σχέση με την ανάγκη που υπάρχει στην Ευρώπη να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Και εδώ έχουμε ένα πολύ καλά σχεδιασμένο εργαλείο που μπορεί να οθήσει τα θέματα αυτά έτσι περαιτέρω και επομένως ε, να ε, δημιουργηθούν πολλά startups από τα διάφορα kicks. Thank you uh, very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Βιδάλ ε, Κουάδρας, σας δίνω το λόγο κύριε Βιδάλ Κουάδρας. Πρόεδρε, ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για την έκθεση του κυρίου Σκίνερ. Θα περιμένω λοιπόν μέχρι ότου παρέμβει πρώτα ο κύριος Σκίνερ και μετά θα μιλήσω. Νόμιζα ότι εγώ ήμουν ο πιο σύντομος παρεμβαίνων, αλλά εσείς ε, με ξεπεράσατε κύριε Δελκαστήγιο. Oh, μιλάμε και για τις δύο εκθέσεις. Πολύ ωραία. Σύντομα λοιπόν θα ήθελα να επισημάνω δύο στοιχεία που είναι ενδιαφέρον θα πιστεύω να ληφθούν υπόψη σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Αφενός πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη επίπτωση και απήχηση όσον αφορά τα ΚΙΚΣ και πρέπει να συνδέονται περισσότερο με την δομή των μέτρων του ορίζοντα 2020 στρατηγικά. Και γι' αυτό θα πρότεινα σε σχέση με την κατάρτιση και εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διασύνδεση με τις δράσεις Marie Curie και με τις δράσεις για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και από την άλλη πλευρά ένα θέμα που πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα και μάλλον ως ορίζοντας εγκάρσια πρωτοβουλία πρέπει να ενταχθεί ώστε να έχει ξεχωριστή, ξεχωριστό άξονα το δυναμικό και η δυνατότητα των start-ups, της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων από μηδενικού σημείου. Αυτό έχει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη τέτοιου είδους επιχειρήσεων, start-ups μέσω του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Ειλικρινά πιστεύω ότι θα έδιναν ένα ευδιάκριτο χαρακτήρα, μια αντανάκλαση της ε, θετικής εικόνας της Ευρώπης σε συσχετισμό με τους τομείς τους πιο επιχειρηματικούς και πιο καινοτόμους της κοινωνίας μας στην Ευρώπη. Και αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ως προς αυτό το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Καινοτομίας και Τεχνολογίας έχει μια ολόκληρη διαδρομή να διανύσει για να είναι αποτελεσματικό και ως ένα άξονα δράσης πρέπει να λάβει αυτή τη, δράση, αυτή τη δραστηριότητα. Έναν ορίζοντα που πρέπει να αναπτύξει πρωτοβουλίες, δεν ξέρω, τώρα άμεσα αμέσως. Εν πάση περιπτώσει, περιπτώσει βραχυπρόθεσμα μέχρι ότου αρχίσει και λειτουργεί και δραστηριοποιείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Με τροπολογίες αυτό θα προτείνω. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Οντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θυμάμαι Όταν είχαμε δουλέψει στην ενδιάμεση επισκόπηση του 7ου προγράμματος, οι αξιολογητές είχαν ζητήσει να σταματήσουμε τη δημιουργία επιπλέον δομών στον τομέα της έρευνας. Εγώ νομίζω ότι θα είμαστε πολύ σόφρονες όταν ε, προτείνουμε ναι, ε, πολλαπλασιασμό των ε, δομών όσον αφορά την γνώση και ε, τη διάχυση της πληροφόρησης και της γνώσης βεβαίως. Εγώ ε, συμφωνώ να μπορεί η βασική έρευνα ε, να μετουσιωθεί σε γνώση και να τελικά να οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη. Δεν έχω τίποτα εναντίον αυτού, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πρώτον να μην δημιουργήσουμε υπερβολικά πολλές δομές Αναρωτιέμαι επίσης την χρήση και το, την ε, ε, χρησιμότητα, την ωφέλεια ε, επιπλέον δομών. Μου εξήγησαν ότι αυτό θα έχει σαν στόχο την εξέβρεση ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να δημιουργήσουμε μια σειρά δομών, δηλαδή πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο, ελεγκτή λογιστή κτλ γιατί εμένα με τρομοκρατούν όλα αυτά. Ε, γιατί ξέρετε έχουμε περάσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με αυτές τις εκστρατείες ε, επικοινωνίας που δεν οδηγούν πουθενά τελικά. Επίσης όλες αυτές οι κοινωνίες ε, οι οποίες ε, δημιουργούνται ε, καλό είναι αλλά θα ήθελα να βεβαιωθώ, να μου δώσουν τι δηλαδή, τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι το ΕΙΟΤΑΤΑΦ θα, θα είναι ακριβώς ευρωπαϊκό γιατί ξέρετε εμείς δημιουργήσαμε δεκάδες υπηρεσίες με ε, δεκάδες συμβούλια των οποίων προεδρεύουν διευθυντές οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και ότι δεν ε, εξαρτώνται από κανέναν. Εγώ θα ήθελα να είμαι σίγουρη, σίγουρος ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι πολιτικώς εξαρτώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος και ο διευθυντής θα πρέπει να ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και επομένως ε, θα, θα πρέπει να έχουν και την σαφή δέσμευση να μην ξεφεύγουν από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και να προσπαθούν να τους επιτύχουν. Εάν καταλαβαίνω καλά το καταστατικό του ΕΙΤΑΦ ΕΕ, υπάρχει μια διευθυντική επιτροπή, ένα κομιτέ directeur το οποίο έχει όλες τις εξουσίες στα χέρια του. Συμφωνώ με την αναθεώρηση του καταστατικού του ΕΙΤΑΦ ΕΕ, ε, και στα πλαίσια αυτά να ξαναδούμε την κατάσταση και να βεβαιωθούμε ότι και αυτή η δομή θα είναι πραγματικά υπό την έγκαιρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, καταλαβαίνω βεβαίως ε, τη θέση της κυρίας Ματίας σε σχέση με το Στρασβούργο, αλλά ξέρετε, είναι λίγο χονδροειδές Καταλαβαίνω, κυρία Ματίας, ε, ότι θέλετε το καλύτερο για το Στρασβούργο, έχετε κάθε συμφέρον, αλλά νομίζω ότι η περιφέρεια του Στρασβούργου, ο Δήμαρχος και οι υπόλοιποι μπορούν να αποφασίσουν για το τι είναι καλύτερο για το Στρασβούργο. Ε, εγώ νομίζω ότι αυτό ότι θα πρέπει να έχουμε σύντομα μια πολιτική συζήτηση για τις έδρες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μονάχα για το Στρασβούργο, ε, ε, να λάβουμε υπόψη μας και πολλά άλλα στοιχεία, όπως ας πούμε είναι η σπανιότητα των δημοσίων πόρων, όπως ας πούμε οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Πολλά στοιχεία θα πρέπει ε, να ληφθούν υπόψη για αυτό το θέμα. αυτή η δομή για την έρευνα θα πρέπει να γίνει σωστά, άσχετα από το ε, τι πρέπει να κάνουμε με το Στρασβούργο και αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, τα κτίρια του Στρασβούργου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και συμφωνώ και με την άποψή σας σε πολλά θέματα και είμαι βέβαιος ότι η κυρία Ματίας έκανε μία πρόταση με πιο επικοδομητικό τρόπο όπως την έκανα εγώ από ό,τι έκανα εγώ όταν απάντησα. Ήσασταν όλοι πολύ καλοί και έχω λίγο χρόνο στη διάθεσή μου για αυτό το τμήμα της συζήτησης και θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα στους δύο εισηγητές να πούν ε, οτιδήποτε επιπλέον μπορεί να θέλουν να προσθέσουν. Κυρία Ματίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα. Να ξεκινήσω με τον κύριο Τσουκαλά. Συμφωνώ πολύ με τα όσα είπατε κύριο Τσουκαλά. Ο κύριος Γιώχανσεν στη συνέχεια και με αυτά που άκουσα από εσά συμφωνώ και θα το δείτε αυτό διότι η πρόταση φαίνεται ότι έχει διαφορετικές διαδικασίες για την επιλογή των ΚΙΚΣ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κλειστές αυτές οι έξι θεματικές ενότητες, διότι μιλάμε για ένα διάστημα 7 ετών. Αυτό είναι μεγάλο χρονικό διάστημα και πολλά μπορούν να αλλάξουν Δεν θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να είναι κλειστός ο κατάλογος εκ των προτέρων. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν ε, θα ξεκινήσει το 2013 θα δούμε τι έχουμε, θα δούμε από εκεί και πέρα και πόσα ε, θα δημιουργηθούν επί τη βάση των προτεραιοτήτων που θα θεωρήσουμε ότι είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε. Υπήρξε κάποια ανησυχία για τον ρόλο του οποίο, τον οποίο θα διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας σε θέματα παιδείας. Δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για ένα Ινστιτούτο το οποίο θα χρηματοδοτήσει μόνο έναν κατάλογο του τριγώνου έρευνας, καινοτομίας και παιδείας, αλλά τα πανεπιστήμια με κοινοτόμα προγράμματα τα οποία θα μπορέσουν να εκπαιδεύσουν νέους της Ευρώπης ε, και εντός αυτών των προγραμμάτων ε, θα πρέπει να τηρούνται κάποια στοιχεία. Δεν θα πρέπει να τηρούνται όλα όσα εμφανίζονται σε αυτό το, το τρίπτυχο τα κίξ ε, δεν θα πρέπει να είναι όλα το ίδιου με σου. Δεν υπάρχει ένα μέγεθο και ένα προπολογισμό για το καθένα. Το καθένα θα έχει διαφορετικό μέγεθο και διαφορετικό προπολογισμό, ο οποίο θα καθορίζεται ανάλογα και μετά όσα έχουμε στη διάθεσή μα. Στη συνέχεια, ο κύριο Τσίτσεστερ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι αρκετά απεπισμένη για τις δυνατότητες που έχει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Τεχνοτομίας. Μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση επαόριστον άμα θέλετε, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό το κέντρο είναι αυτό το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε την Ευρώπη της καινοτομία και της γνώσης. Συμφωνώ και με τα όσα ακούσαμε την κυρία Πιλάρτε Καστίγιο για τα startups και στα όσα είπε ο κύριος Ντοή, συγγνώμη, για διάφορα ζητήματα. Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε εκ νέου νέους υποδομής και συμφωνώ και για την εμπειρία και τα όσα ακούστηκαν. Τέλος, για το Στρασβούργο. Προφανώς εγώ δεν αναφερόμουν στο Στρασβούργο ως πόλη, Αναφερόμουν στα κτίρια, τα οποία είναι δικά μα. ανήκουν σε όλους τους Ευρωπαίους και νομίζω ότι η πρότασή μου είναι επικοδομητική. Δεν χρειάζεται να στερήσουμε τίποτα ούτε από τη Γαλλία ούτε από το Στρασβούργο. Θέλουμε να προσθέσουμε κάτι, ίσα ίσα να του προσφέρουμε κάτι του Στρασβούργου. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να προτείνουμε συγκεκριμένε προτάσει. Λένε οι συνάδελφοι ότι δεν είναι ο κατάλληλο χώρο για να υπάρχει και αυτή η πρόταση. Και πότε είναι ε, και πού ο κατάλληλο χώρο. Δεν θέλουμε να στερήσουμε τίποτα από το Στρασβούργο, επαναλαμβάνω. Θέλουμε να του δώσουμε κάτι επιπλέον, πλήρη απασχόληση αν θέλετε. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Διότι το κτίριο και η πόλη είναι πολύ ωραία ε, και δεν χρειάζεται μόνο να πηγαίνουμε 3,5 μέρε το μήνα. Ο κύριο Λάμπερτ. Δεν θα απαντήσω σε όλα τα σχόλια. Είμαστε εδώ για να συμφωνούμε και να διαφωνούμε, αλλά παρόλα αυτά ούτως ή άλλως βλέπω, θα δω τις τροπολογίες. Λοιπόν, ε, ε, Λάμπερτ, περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία ε, τις τροπολογίες σου γιατί ίσως δώσεις κάποιες ιδέες σχετικά με την καλύτερη διασύνδεση κάποιων ιδεών. Εάν το επιτύχεις πραγματικά θα είμαι πάρα πολύ ανοιχτό μυαλός με όσα θα κομίσεις και θα τα λάβω υπόψη μου. Σε αυτά που είπε ο Ζαν Πιέρ ε, λες ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν ε, νέες ε, νέες ε, υπηρεσίες ε, και ε, από την άλλη πλευρά μου αναφέρεσε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογία Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα έχουμε θα έχω μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Τεχνολογίας, τον διευθυντή μάλλον. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ ανοιχτό πνεύμα και επομένως νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο τρόπο θα έχουμε καλύτερη ευελιξία του οργάνου, ε, ε, καν, ταυτόχρονα όμως <laughs> να είναι σαφές ότι ακολουθεί ε, την ευρωπαϊκή οδό. Εδώ συμφωνώ μαζί σου. Εκεί όμως που είμαι λίγο, με αφήνει σκεπτικό είναι το εξή. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε την ευκαιρία να αρχίσουμε να σκοτώνουμε κατά κάποιο τρόπο την Bird η η οποία πλέον δεν έχει και έννοια να παραμείνει ζωντανή από τη στιγμή που έχουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ναι, είναι γεγονός ότι θα πρέπει λίγο ε, να νοικοκυρέψουμε την κατάσταση όσον αφορά ε, όλα αυτά τα προγράμματα, όλους αυτούς τους οργανισμούς, όλα ε, αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολλά και είναι γεγονός ότι για τον ορίζοντα 2020 έχουμε διάφορους οργανισμούς που θέλουν να δουλέψουν ε, σαν σιλό. Ξέρετε πώς είναι τα σιλό που θέλει ο καθένας να έχει το δικό του κομμάτι του προγράμματος, το δικό του κομμάτι της ε, χρηματοδότησης. Ε, εν πάση περιπτώσει, εάν εδώ στην Ήτρε υπάρχει και προκύψει πλειοψηφία η οποία να λέει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε, να, να, να κλείσουμε ε, κάποιες ε, υπηρεσίες, ναι, γιατί όχι. Αυτό που θέλουμε πάντως ε, σίγουρα είναι στην ενδιάμεση επισκόπηση του ορίζοντα 2020 να είμαστε πάρα πολύ ε, αυστηρή, να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα χρήματα με λιγότερε δομέ. Εγώ δεν έχω κανένα ταμπού ε, και καμία προκατάληψη όσον αφορά το θέμα αυτό. Με το ίδιο επικριτικό βλέμμα βλέπω και εγώ όλη αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την συζήτησή μα για αυτή ε, την κοινή μα συζήτηση. Θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί πρέπει να φύγω, γιατί ε, έχουμε ανταλλαγή απόψεων επί άλλης εκθέσεώς μου σε μια άλλη ε, επιτροπή. Σίγουρα θα μου πούν ε, τι είπατε. ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως τελειώσαμε αυτό το κομμάτι, οπότε μη σας απασχολεί. Σας ευχαριστώ πάντως όλους που είσαστε εδώ, που μιλήσατε σεβόμενοι το χρόνο σας και ε, να καλέσω τον κύριο Σκίνερ να ξεκινήσει ε, για το τρίτο μπλοκ. Δεν το κάνω επίτηδες, πρέπει να φύγω. Δεν το κάνω για σένα. Ε, δεν προσβάλλομαι. Ξέρεις ότι θα μπορούσα να προσβληθώ, αλλά δεν θα προσβληθώ. Λοιπόν, Έχουμε εδώ το πακέτο 2020 και ε, όλο αυτό το πακέτο δίνει την δυνατότητα στους ερευνητές, μάλλον δίνει νέες δυνατότητες στους ερευνητές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η πυρηνική έρευνα ε, και η πυρηνική φυσική. Δεν αφορά βεβαίω την ίδια την πυρηνική ενέργεια ε, και για το κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί, θα επιλεγεί από τα κράτη-μέλη για να χρησιμοποιηθεί ε, απλώς είναι μία μορφή επιστήμης ε, που θα πρέπει να μελετηθεί. Ξέρω ότι υπάρχουν μέλη της Επιτροπής ε, που δεν θέλουν καθόλου αυτήν την ιδέα και δεν καλωσορίζουν το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας μετά κυρίως από το επεισόδιο της προηγούμενης χρονιάς με τον στη Πιστεύω λοιπόν ότι εξ αρχή θα πρέπει να κάνουμε κάποιε βασικέ, να πάρουμε κάποιες βασικές αποφάσεις όσον αφορά την ε, επιστήμη. Ε, επίσης, ε, όσον αφορά την νομική βάση, είναι γεγονός ότι δεν έχουμε ε, την ίδια δυνατότητα αποδοχής και τροπολογίας, αλλά πιστεύω ότι οποτεδήποτε πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υποβάλουμε τροπολογία ή άποψη, θα πρέπει να το κάνουμε. Επίσης, να πω, στο να πω ότι στο Κοινοβούλιο είχα πάρα πολύ καλή συζήτηση και συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές. Όλοι προσπάθησαν να φέρουν κάτι νέο στη συζήτηση αυτή. Ε, εγώ λοιπόν που προέρχομαι και από μια άλλη επιτροπή είναι χρήσιμο να ασχολούμαι στην επιτροπή εδώ με κάτι ενδιαφέρον και να βλέπω ότι μπορούμε να κάνουμε καλή συζήτηση χωρίς όμως ε, απαραίτητα να συμφωνούμε απαραίτητα. Υπάρχουν ε, μέτρα cross-cutting και στην ε, περίπτωση αυτή ε, και εδώ ας πούμε συμπεριλαμβάνω και την διαδικασία απλούστευσης. Η μείωση του διοικητικού άχθους είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και τους ε, εισηγητές, τους εισηγητές, γιατί πάντα μου έδειξαν και νέους τρόπους για να αντιμετωπίσω κάποια θέματα. Επίσης, όσον αφορά ε, τους νέους ερευνητές ε, και τις μικρές επιχειρήσεις, ε, αυτοί αντιμετωπίζουν πολύ συχνά προβλήματα όσον αφορά την βαριά γραφειοκρατία, γιατί δεν έχουν την ίδια διοικητική προετοιμασία με τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις κυρίως δε τώρα που οι οικονομικές συνθήκες είναι πιο δύσκολες. Διεθνή συνεργασία, θεωρώ ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον. Όσον αφορά ας πούμε το ατύχημα στην Φουκουσίμα ε, θα πρέπει στενά να συνεργαστούν όλοι ε, έτσι ώστε να αποφευθούν παρόμοια ατυχήματα εις το μέλλον και νομίζω ότι μέσω αυτής της έκθεσης ε, και μέσω του ορίζοντα 2020 μπορούμε να δούμε να, επιτύχουμε βελτιώσεις. Πρόσφατα ο πρόεδρος Βαν Ρόμποϊ είπε ότι θα πρέπει να αυξηθούν ε, σε παγκόσμιο επίπεδο τα ε, ε, τα επίπεδα της ατομικής πυρηνικής ασφάλειας. Ναι, βεβαίως αυτό θα γίνει και παντού. Ε, έχουμε νέες χώρες και πολλές χώρες οι οποίες θέλουν να έχουν πλέον χρήση και παραγωγή και χρήση της ε, πυρηνικής ε, ενέργειας. Άρα θα πρέπει να προταθούν στην Ευρώπη διάφορα πρότυπα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και στην Ευρώπη αλλά και αλλού. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, στην, ε, στον τομέα της έρευνας για την πυρηνική ενέργεια. Ε, τα τεστ αντοχής που έγιναν πρόσφατα μας έδωσαν πολλά στοιχεία όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια. Υπογράμμασα, υπογράμμισα ότι η προστασία των εργαζόμενων, η προστασία όλων όσων ασχολούνται με το θέμα έχει, είναι πάρα πολύ σημαντική. Τρίτον, ή τα και το μέλλον της ε, ε, τήξης, της σύνδεξης. Όλα αυτά αναφέρονται εδώ. Ξέρετε ε, ότι στις προτάσεις της η Επιτροπή δεν έχει συμπεριλάβει το ΙΤΑ και ε, αυτό μπορεί να είναι σημαντικό θέμα, αλλά βεβαίως ε, πιστεύω ότι ε, πέρα από τις συζητήσεις που θα γίνουν στο Συμβούλιο, θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει την άποψή του σαφώς για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να, να, να υπάρξει η χρηματοδότηση του ΙΤΕΡ, ενδεχομένως μέσω των πολιετών χρηματοδοτικών προοπτικών. και βεβαίως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να δηλώσει σαφώς και κατηγορηματικά ότι θα χρηματοδοτήσει το μέλλον της σύνδεξης, ότι θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί το, να ε, το ε, ίτερ. Περιμένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει την θέση της. Ε, και εν πάση περιπτώσει το ίτερο ό,τι και να θέλει να πει κανείς ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι μια μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να την αφήσουμε να χαθεί. Επίσης θα πρέπει να στηριχτεί η έρευνα για την σύνδεξη. Ε, ε, δεν θα πρέπει επομένως να σταματήσει και η λειτουργία του JET και η λειτουργία του ITER. Ε, Στον ορίζοντα 2020 δεν έχει καμία έννοια να αρχίσουμε να έχουμε κενά, γιατί εάν αρχίσουν να φεύγουν τα καλά μυαλά, τότε θα είναι το χειρότερο για το ΙΤΕΡ. Όσον αφορά την ε, χρηματοδότηση, έχουν ε, ε, καθοριστεί τα, οι χρηματοδοτήσεις για την σύνδεξη και βλέπουμε ότι έχουμε μια πολύ μικρή αύξηση σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να βοηθηθούν όλα τα κέντρα τα οποία θα πρέπει να σταματήσουν την λειτουργία τους, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ε, όσον αφορά τον προϋπολογισμό δεν έχουμε ακόμα τα τελικά στοιχεία. Ελπίζω ότι θα υπάρξουν και μελλοντικέ συζητήσεις με τους συναδέλφους έτσι ώστε να ε, καταλήξουμε σε ένα λογικό συνολικό προϋπολογισμό ο οποίος θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις ανάγκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, τον συνάδελφο Σκίνερ. Ο κύριος Μπρετζίνα, μάλλον ο μόνος παρόν σκιώδης εισηγητής είναι, που είναι παρόν. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή την πολύ ισορροπημένη έκθεση. Ε, ο εισηγητής υπογραμμίζει ε, τα ευρωπαϊκά στρατηγικά προγράμματα τα οποία έχουν ε, ήδη ε, οριστεί και αναφέρεται επίσης και στις πρωτοβουλίες που αφορούν την βιώσιμη πυρηνική σύνδεξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό βεβαίως να υπάρχει ο απαραίτητος βαθμός επιστημονικής ετοιμότητας αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι τα κράτη-μέλη είτε χρησιμοποιούν είτε δεν χρησιμοποιούν την πυρηνική ενέργεια, όμως η επιστήμη ε, θα πρέπει να συνεχίσει την έρευνα για την ε, πυρηνική ενέργεια έτσι ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ε, στον τομέα αυτό. Πρέπει να, έχουμε, να είμαστε εμπειρογνώμονες στο θέμα αυτό έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα σε αφορά την μελλοντική μας ανταγωνιστικότητα. Δεν συμμερίζομαι απόλυτα την ιδέα ότι είναι δυνατόν σε μικρό χρονικό διάστημα να επιτύχουμε συμφωνία για το ΙΤΕΡ. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα λέγοντας ότι όσον αφορά αυτήν την ζωτική για το μέλλον της Ευρώπης τεχνολογία θα πρέπει να επενδύσουμε. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να στηρίξουμε και άλλα συμπληρωματικά προγράμματα τα οποία αφορούν την ε, πυρηνική σύνδεξη και να πούμε ότι και στα πλαίσια του πολιετούς ε, χρηματοδοτικού πλαισίου θα πρέπει να γίνει αναφορά στην ε, χρηματοδότηση της πυρηνικής ενέργειας. Ε, όσον αφορά τον όγκο των διοικητικών ε, ε, εξόδων που είναι 13,5% στο έγγραφο αυτό, συνήθως είναι 8% και λαμβάνοντας υπόψη και ότι ο προϋπολογισμός γενικά ε, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος, προτείνω η, η ε, η οικονομία ε, που θα πρέπει να γίνει στα ε, διοικητικά έξοδα να χρησιμοποιηθεί για την έρευνα για την πυρηνική σύνταξη. Επίσης θα ήθελα μεγαλύτερη αναφορά στους αντιδραστήρες τέταρτης γενεάς που θα πρέπει να οικοδομηθούν γιατί πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δύο λεπτά ε, θα έχουν στη διάθεσή τους ε, οι σκιώδεις. Ο κύριος Μπρετσίνα σεβάστηκε το χρόνο αυτό. Επόμενος ομιλητής τώρα. Κρότσμαν, ευχαριστώ πολύ. Ο καθηγητής Παναγιώτοφ δεν μπορεί να παρασύσει συζήτηση. Θα σας διαβιβάσω κάποιες παρατηρήσεις του σε σχέση με την έκθεση του κυρίου Σκίνερ ως γεώδος εισηγητή, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Ο στρατηγικός ορίζοντας 2020 στοχεύει να δώσει τη βέλτιστη συμμετοχή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των, που αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας. Μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και κατάτησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας συμπληρώνοντας τον χρονορίζοντα 2020 έχουμε υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ζωτικό ρόλο μακροπρόθεσμα η έρευνα. Αν τα κράτη-μέλη αποφασίσουν να συνεχίσουν την πυρηνική ενέργεια, θα πρέπει τότε να έχουμε ένα φιλόδοξο πλαίσιο για την έρευνα, την κατάρτιση, για να διασφαλιστεί η συνιστόσα της ασφάλειας ε, της εκμετάλλευσης πυρηνικής ενέργειας, βέλτιστη χρήση των πόρων και της πραγματογνωμοσύνης ε, και προαγωγή περαιτέρω υπεροχής και βέλτιστης ε, ε, δραστηριότητας και δράσης και διάχυση και διάδοση των γνώσεων στον τομέα. Είναι σημαντική αυτή η συνιστόσα για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και της ε, εκμετάλλευσης του άνθρακα. Θα πρέπει εδώ να δούμε ότι υπάρχει ένα σημαντικό ρόλο, ένα σημαντικό εργαλείο με συγχωρείτε για την έρευνα και την ανάπτυξη στο ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει να στοχεύουμε στο να έχουμε μια πιο αποτελεσματική έρευνα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους τα κράτη-μέλη για την έρευνα, τη δημιουργία μιας βάσης ε, τη δημιουργία της βάσης γνώσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς επίσης και της ασφάλειας, την, της αντιμετώπισης των θεμάτων ακτινοβολίας ε, χάρη της ασφάλειας και την αντιμετώπιση όλων των άλλων προκλήσεων. Διεθνή συνεργασία μέσω των ευρωπαϊκών σημαντικών στατηγικών εταίρων έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την συνέργεια και συντονισμό δράσεων για να διασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και προδιαγραφών στην Ευρώπη και παγκόσμια όσον αφορά την συνεργασία σε αυτόν τον τομέα. Να βελτιωθεί η συμμετοχή τρίτων κρατών στην συμμετοχή στην έρευνα μέσω μιας δυνατότητας να βοηθήσουμε από τη διεθνή κοινότητα αυτές τις χώρες και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι προπομπός όσον αφορά τις πτυχές αυτές της έρευνας και της κατάρτισης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Μάλιστα σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σε κάποια θέματα με θετικό πνεύμα για την έκθεση του κυρίου Σκίνερ. Για παράδειγμα, όσον αφορά την αντίστασή του, την αντίθεσή του για την χρηματοδότηση του ΙΤΕΡ, για παράδειγμα, εκτός του ε, πολιετούς ε, πλαισίου στη, σε σχέση με την έρευνα. Εγώ συμμερίζομαι αυτή την προσέγγιση του για την αιμονή του, για την σημασία που έχει η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για να μπορέσουμε να εξαγάγουμε τις δικές μας προδιαγραφές που είναι πολύ υψηλέ για την ασφάλεια και να προσφέρουμε τη γνώση μας και την ευρύτατη πείρα μας σε αυτόν τον τομέα. Και επίσης το μέλημα να βελτιωθούν οι όροι εργασίας για εκείνους που βρίσκονται σε άμεση επαφή για λόγους επαγγελματικούς με υλικό που έχει έντονη ακτινοβολία, ραδιοπυρηνικό υλικό και να συνεισφέρουμε να μην απολέσει η Ευρώπη την υπεροχή της και το ανθρώπινο δυναμικό της όσον αφορά αυτόν τον τομέα της πυρηνικής της ατομικής ενέργειας και να μπορέσει και να προσελκύσει και εξοκοινωτικούς ειδικού και επαΐοντες. Φυσικά το σύστημά μας ε, είναι ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο παγκόσμια. Το τελικό μου σχόλιο, Πρόεδρε, για το σύνολο της δέσμης μέτρων που εξετάσαμε απόψε για τον ορίζοντα 2020, το σύστημα της βελτίωσης για να αντανακλά πιο αποτελεσματικά ένα μέλημα, μια ανησυχία που όλοι συμμεριζόμαστε. Να υπάρξει μια εκμετάλλευση πιο αποτελεσματική των ευρωπαϊκών κονδυλίων Γι' αυτό είναι, σπουδαίο, είναι ιδιαίτερη σπουδαιότητα να υπάρχει καλή διάχυση των στοιχείων και καλή γνώση των στοιχείων αυτών των προγραμμάτων. Να υπάρχει ένα διαφανές πλαίσιο και να είναι το δυνατόν μικρότερο το γραφειοκρατικό βάρος και η προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να βελτιώσουμε ένα από τα μεγαλύτερα χάσματα και ελλείψεις σε σχέση με τους πιο ισχυρούς ανταγωνιστές μας που είναι το πέρασμα, το βήμα από τη γνώση στην παραγωγή προϊόντων, εξειδικευμένων προϊόντων. Ο κύριος Κίνερ τόνιζε το ότι υπάρχει ανάγκη το σύστημα έρευνας να αφορά πρακτικά αποτελέσματα, χειροπιαστά αποτελέσματα στα προϊόντα. Συμφωνώ μαζί του. Όμως για να μπορέσουμε να περάσουμε από την άλλη πλευρά στην, από τη βελτίωση των γνώσεων σε, σε παραγωγή προϊόντων πρώτα πρέπει να παραγάγουμε γνώση. Αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντικό, η σημαντική συνιστόσα της έρευνας και γι' αυτό πρέπει να είναι σαφές ότι οι δύο πτυχές είναι συμπληρωματικές, αλληλοσυμπληρώνονται ταυτόχρονα. Ε, Ευχαριστώ. πολύ. Ο κύριος ε, Χέλμερ. Προτελευταίος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία του. Θα συμφωνήσω για πρώτη φορά πλήρως με τον κύριο Σκίνερ. Τρομερό. Αναφέρθηκε στη Φουκουσίμα και στο γεγονός ότι κάποιοι συνάδελφοι ε, στην Επιτροπή έχουν επιφυλάξει όσον αφορά την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας. Να σας πω ότι ε, ήμουν σε μια συζήτηση που έγινε για το θέμα αυτό στην, ε, στο, σε ένα Βρετανικό Πανεπιστήμιο και πραγματικά κάνοντας μια έρευνα εν ώψη αυτής της συζήτησης ε, εξεπλάγινα από το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ασφαλής η πυρηνική ενέργεια, πολύ πιο ασφαλής από την υδροελεκτρική ενέργεια. Δηλαδή πεθαίνουν ε, ένα σωρό άνθρωποι στα υδροελεκτρικούς σταθμούς και δεν το μαθαίνει κανένας. Ε, πεθαίνουν ε, τρεις άνθρωποι στη Φουκουσίμα σε πυρηνικό αντιδραστήρα. Όλος ο κόσμος παθαίνει κρίση. Η Γερμανία σταματάει το πυρηνικό της πρόγραμμα και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί όσον αφορά αυτό το θέμα. Βεβαίως θα πρέπει θα έπρεπε να μπορούσαμε να έχουμε εθνικά προγράμματα αλλά αλλά εάν ε, πρέπει να περάσουμε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, α το κάνουμε αν δεν έχουμε άλλο τρόπο. Αυτό ήθελα να πω και συγχαρητήρια, Πίτερ. Ευχαριστώ, κύριε Έλμερ. Ε, τον λόγο έχει ο κύριο Σοντή. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Μερικές παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον εισηγητή για την ποιότητα της έκθεσής του. Ε, βεβαίως ε, έχουμε και το κοινό πρόγραμμα, ε, συγγνώμη, το κοινό κέντρο ε, έρευνας, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό όσον αφορά την έρευνα για την ασφάλεια ενεργητική και παθητική στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Ε, όσον αφορά την έρευνα για την ε, κατάργηση πυρηνικών ε, εγκαταστάσεων και πυρηνικών αντιδραστήρων, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξέρουμε με ποιο τρόπο θα πρέπει να προχωρήσουμε έτσι ώστε να έχουμε τις καλύτερες προδιαγραφές σε όλο τον κόσμο. Δεύτερον, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τις προθεσμίες για τα προγράμματα. Για τα προγράμματα που ολοκληρώνονται δεν υπάρχει ασυνέχεια, αλλά υπάρχει ε, ε, μία ας πούμε ε, ασυνέχεια όσον αφορά το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και το Ευρατόμ γιατί θυμάστε ότι είχε προταθεί ε, η ε, διατηρηθεί για δύο ακόμα χρόνια πριν από το ατύχημα της Φουκουσίμα. Δεν ξέρω πώς σε αυτόν τον κανονισμό μπορούμε να εισάγουμε ε, το ζήτημα αυτό και πώς θα το διασυνδέσουμε και με τον ορίζοντα 2020, γιατί η προθεσμία είναι πενταετής. Ε, πώς θα μπορούσαμε λοιπόν στο κείμενο αυτό ήδη να προβλέψουμε ότι θα υπάρξει επιμήκυση των, πέντε χρόνων έτσι ώστε να ταυτιστεί με τον ορίζοντα 2020 ενδεχομένως ε, μέσα από την εισαγωγή ε, μίας σειράς ή ενός χρονοδιαγράμματος αξιολογήσεων. Τελευταίο σημείο. Γνωρίζετε βεβαίω ότι εμεί γνωμοδότηση κάνουμε. Δεν είναι ότι δεν αποφασίζουμε τίποτα, αλλά βεβαίω το Συμβούλιο αποφασίζει. Μόνο διαβούλευση γίνεται με το Κοινοβούλιο. Ε, γιατί η νομική βάση είναι η συνθήκη Ευρωτόμου που είναι διακυβερνητική. Ε, η εξέλιξη των πραγμάτων, η εξέλιξη της τάση των πολιτών μας οδηγεί στο να πρέπει να κατανοήσουν ε, οι, οι πολιτικοί ταγοί ότι ε, δεν είναι δυνατόν να περνούν όλα αυτά τα χρόνια χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να συμμετέχει με συναπόφαση. Ε, δεν μιλάω για αναθεώρηση των συνθήκων. Μήπως όμως θα μπορούσαμε μέσω εισαγωγής τροπολογίας να δώσουμε μεγαλύτερο ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα έλεγα ας πούμε να έχει ε, συμβουλευτικό ρόλο στην απόφαση και την εξέλιξη του προγράμματος. Γιατί κάθε φορά είναι ιδιαίτερο αγχωτικό το γεγονός ότι ε, το Κοινοβούλιο συζητάει σαν να ήταν σε συναπόφαση, αλλά δεν είναι σε συναπόφαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Μπουτικόφερ, παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο. Ε, Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, δεν ήθελα να παρέμβω. Αλλά μια και ο συνάδελφος Χέρμερ μίλησε για την Γερμανίδα καγκελάριο και δυστυχώς δεν υπάρχει κανείς από την Τσεντεού να την υπερασπιστεί. Θέλω να το κάνω εγώ. Στην κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας πολύ ορθολογικά έδρασε με την απόφαση αυτή. Πολύ ωραία. Και με αυτή τη δήλωση του κυρίου Μπουτκόφερ μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Σμίτς, ο οποίος ε, θα καλύψει τα πάντα για τα διάφορα τμήματα τα οποία συζητήσαμε για το Horizon 2020. Ένα πεντάλεπτο σας δίνουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και καταρχάς να συγχαρώ όλους τους συζηγητές και τους κοιόδης συζηγητές για την δουλειά τους η οποία ήταν πρώτης τάξος. Χαίρομαι που συνεργάζομαι μαζί σας, διότι συζητάμε ένα τεράστιο ποσό χρημάτων και πρόκειται και για μια πρόταση η οποία ε, χρήζει όλης μας της προσοχής. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα-δυο σημεία. Καταρχάς, ε, η δομή του Horizon 2020. από ό,τι διαπιστώνω, οι περισσότεροι από τους εισηγητές και οι σκιώδεις εισηγητές ε, προσυπογράφουν την προτινόμενη δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, υποστηρίζουν το να συνδέσουμε την έρευνα με την καινοτομία και υποστηρίζουν σε γενικές γραμμές την πρότασή μας. Ε, κάποιες ιδέες να αποσυνδέσουμε ε, την προτεραιότητα 6 και να βρίσκεται η ασφάλεια σε διαφορετικό τμήμα δεν μας αρέσει και πάρα πολύ. Για μας είναι πολύ σημαντικό οι κοινωνικές επιστήμες, οι ανθρωπιστικές επιστήμες και η ασφάλεια να βρίσκονται ε, στην ίδια πρόκληση διότι υπάρχει μια σχέση. Αν μιλήσουμε για ασφάλεια στους πολίτες και για την τρομοκρατία υπάρχουν κοινωνικές ε, πτυχές και θα ήταν σφάλμα κατά την άποψή μας να διαχωρίσουμε τα δύο και χαίρομαι ε, που το επεσήμανε και ο κύριος Λάμπερ, ο οποίος είπε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι το θέμα της ε, διεύρυνσης της συμμετοχής και το να διασφαλίσουμε ότι το ορίζον 2020 είναι προς όφελος όλων των κρατών μελών και όχι μόνο μερικών. Κύριε Μπούζεκ, νομίζω εσείς αναφερθήκατε σε αυτό και κάποιος άλλος. Ε, Μα ανησυχεί ιδιαίτερα να υπάρχει διαχωρισμό μεταξύ έρευνα και καινοτομία. Θα θέλαμε το ε, πρόγραμμα να απευθύνεται σε όλε τι χώρε και σε όλε τι περιφέρειες. Γι' αυτό και ακριβώ δεσμευόμαστε για να δημιουργήσουμε αυτή την κλίμακα αριστεία. Και νομίζω ότι στο παρελθόν έχουν γίνει συζητήσει εδώ στην Επιτροπή σα. Ε, και ξέρουμε ότι πρέπει να γίνει πολύ μεγάλο μέρο τη δουλειά μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, διότι αναφερόμαστε στα διαρθρωτικά ταμεία, στην επένδυση στι δυνατότητέ μα, σε νέα πανεπιστήμια, σε εξυγχρονισμό εξοπλισμού και ούτε καθεξής, αλλά το ορίζον 2020 ε, θα περιλαμβάνει και αρκετέ δραστηριότητε ε, για να διασφαλίσει ότι θα γίνει πράγματι αυτή η διεύνηση. Και κατά την άποψή μα, αυτέ οι δραστηριότητε δεν θα πρέπει να βρίσκονται στον πρώτο πυλώνα τη αριστεία, αλλά θα πρέπει να βρίσκονται ε, στην πρόκληση υπαριθμών 6 για τι προκλήσει τη κοινωνία, όπω είχαμε προτείνει αρχικώ. Κύριε Μπούζεκ, αναφερθήκαμε στην κλίμακα αριστεία. Περιμένουμε και την πρόταση του κυρίου Ρόλ για την αδελφοποίηση της αριστείας ε, και χαιρόμαστε που δεν είμαστε οι μόνοι που ενδιαφερόμαστε για το θέμα αυτό. Πριν από κάποιες εβδομάδες ακούσαμε και τον πρόεδρο της κοινότητας Max Planck, ο οποίος ήταν παρόν ε, στην διπλανή αίθουσα που ήθελε και αυτός να αναλάβει τις ε, ευθύνε του και ήθελε να υπάρχουν κάποιες κοινέ δραστηριότητες με ομάδες από διάφορα τμήματα της Ευρώπης, ώστε κάποια τμήματα αριστείας, κάποιες δυνητικές πτυχές της αριστείας να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στο σύστημα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ετοιμάζουμε και σχετικό έγγραφο επί του ζητήματος, διότι για μας είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό και πραγματικά πρέπει να πω στην κυρία Μαντουρέλ και στην κυρία Καρβάγιο ότι αυτό βρίσκεται στις προτεραιότητές μας σε πολύ ψηλή θέση. Γι' αυτό λοιπόν θα βεβαιωθούμε ότι θα υπάρξει και αποτέλεσμα. Τρίτη παρατήρηση, θέματα προϋπολογισμού. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αρκετά ποσοστά τα οποία αναφέρονται στην πρόταση της κυρίας Μαντουρέλ για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Εμείς είμαστε υπέρ ε, του να υπάρχει ακόμα κάποια ευελιξία στον προϋπολογισμό, διότι ε, αρκετές φορές είτε πρόκειται για τις τρελές αγελάδες, σπογγόδια κεφαλοπάθεια ή οτιδήποτε άλλο, αν έχουμε διαθέσει ποσά μέχρι το τελευταίο σετ του ευρώ, είναι πολύ δύσκολο να αποδεσμεύσουμε κονδύλια για να αντιμετωπίσουμε την ε, σπογγόδια ε, κεφαλοπάθεια και την γρήπη των πτηνών. Ε, πρέπει να υπάρχουν κάποια κονδύλια στην άκρη για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες κατεπήγουσες ανάγκες. Τέταρτη παρατήρηση, η οποία έχει μεγάλη σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Αρκετοί από σας αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό. Θέλουμε η βιομηχανία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμπεριληφθούν στο ε, πρόγραμμα όσο το δυνατόν περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν. Ε, κάποιοι από εσά χαιρέτησαν την προσέγγιση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, το ε, πρόγραμμα SBIR, το οποίο έχουμε προτείνει και εδώ υπάρχει ένα στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πώ θα καθορίσουμε την ανοιχτή πρόσβαση, διότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ τη μόδα η ανοιχτή πρόσβαση για τι διάφορε δημοσιεύσει, αλλά δεν είναι το ίδιο με την ε, ανοιχτή πρόσβαση για τη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα. Ορισμένε φορέ το να επιβάλλουμε την ανοιχτή πρόσβαση ω γενικό κανόνα για την έρευνα ε, θα σημαίνει ότι ο κλάδος, η βιομηχανία, η οποία πολλές φορές χρηματοδοτεί, δεν θα συμμετέχει και δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ναι λοιπόν στην ανοιχτή πρόσβαση, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς ως προς τα ποια κριτήρια θα πρέπει να ισχύσουν και ποιες προϋποθέσεις. Και κάποιοι από εσά το επεσήμαναν. Ε, πέμπτη παρατήρηση, απλούστευση. Η κυρία Νούιμπλερ ανέφερε πόσο σημαντική είναι αυτή η απλούστευση και νομίζω ότι αυτό είναι το ήπιο τμήμα του ορίζοντα 2020, η απλούστευση. Μας ανησυχεί λίγο όταν ακούμε οι ιστορίες, ε, το να υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά χρηματοδότησης για διάφορες κατηγορίες. Θυμάμαι πολύ καλά την παρέμβαση του εκπροσώπου του Ελεκτικού Συνεδρίου, του κύριου Μπάλκο, σε μία ακρόαση του ΕΛΚ ε, πρόσφατα. Μας είπε, αν θέλετε να πλουστεύσετε, κρατήστε τα πράγματα απλά με ένα ποσοστό χρηματοδότησης το οποίο θα ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες. Ένα ποσοστό για τις ε, έμεσες χρηματοδοτήσεις και όχι άλλες ε, καταγραφές. Ε, το κατέστησε σαφέ. Να μην υπάρχουν πλέον διαφοροποιημένα ποσοστά, εάν θέλουμε να είναι απλά τα πράγματα. Το ξέρω ότι θα προκύψει αύριο στη συνεδρίαση με τον κύριο Έλερ, ο οποίο θέλει να επανέλθει στα όσα είχαμε στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο αυτή τη στιγμή, δηλαδή διαφοροποιημένα ποσοστά χρηματοδότηση, σα προειδοποιώ, αυτό σα σημαίνει ότι θα έχουμε τεράστια προβλήματα και ε, θα είναι ε, από πάνω μας ε, να κρέμεται ως δαμόκλειο ε, σπάθη ε, το ελεκτικό συνέδριο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν θέλουμε να έχετε διαφοροποιημένο ποσοστό χρηματοδότηση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αυτέ οι επιχειρήσει έχουν τόσο μεγάλε δοκιμάσει προσωπικού που τη μία μέρα είναι μικρομεσαίε επιχειρήσει και την άλλη μέρα δεν είναι γιατί προσλαμβάνουν προσωπικό. Αυτό θα σημαίνει ότι θα εμπίπτουν σε διαφορετικέ κατηγορίε χρηματοδότηση με όλα τα προβλήματα τα οποία συνοδεύουν όλο αυτό το τμήμα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ε, προσέξετε, σα κάνω έκκληση να κρατήσετε τα πράγματα απλά. Τώρα, για την έκθεση της κυρίας Σκίνερ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που επισημαίνεται τη σημασία της πυρηνικής ασφάλειας Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και για την υποστήριξη του προγράμματο ΣΥΤΕΡ και το γεγονό ότι επισημαίνεται ότι χρειάζεται διεθνή συνεργασία και ακόμα και για αυτού που ίσω δεν είναι υπέρ τη πυρηνική ενέργεια, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι υπάρχουν αρκετοί πυρηνικοί αντιδραστήρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, οι οποίοι θα πρέπει να παροπλιστούν και για του οποίου χρειάζεται εμπειρογνωμοσύνη για τα επόμενα 20 χρόνια. Και επιπλέον, εάν υπάρχουν αρκετέ χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, εξοπλίζονται πυρηνικά και ε, λαμβάνουν πυρηνική ενέργεια, τότε θα πρέπει να έχουμε ε, αρκετά στοιχεία ε, ασφάλειας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη και για θέματα ασφαλείας πυρηνικής ενέργειας, αλλά και για ε, εμπειρογνωμοσύνη για τον παροπλισμό των πυρηνικών αντιδραστήρων. Και χαίρομαι κύριε Σκίνερ που τα αναφέρετε στην έκθεσή σας αυτά. Ε, υπάρχουν κάποια άλλα σχόλια. Κύριε Οντή, είπατε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός πταετούς ε, προγράμματος ε, πλαίσιο και ε, μιας Ευρατόμ. Νομίζω ότι ήγηκε η ώρα να γίνει η παράταση της πρότασης Ευρατόμ, όπως το κάναμε και στο παρελθόν, γίνονται γέρος αυτά όλα και χαίρομαι για την πρότασή σας και πρέπει να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι θεσμικό για την Ευρατόμ δεν υπάρχουν οι ίδιες δυνατότητες από πλευρά Κοινοβουλίου όπω το Συμβούλιο, εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάντα το θέτουμε το θέμα προς συζήτηση της Ευρατόμ εδώ σε εσά και λαμβάνουμε υπόψη τα όσα μας προτείνεται παρά το γεγονός ότι βάσει της συνθήκης δεν έχετε τα ίδια προνόμια και δικαιώματα στο θέμα αυτό όπως και το Συμβούλιο. Μακρηγόρησα να σας ευχαριστήσω όλους για την εξαιρετική συνεργασία και ελπίζω να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όπως και μέχρι τώρα προς όφελος ε, και προς χάρη του ορίζοντα 2020 της επιστήμης και της έρευνας και των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ και εγώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα έχουμε τρεις από τους πέντε συγχυτές παρόντες και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για πολύ λίγο στον καθένα για να απαντήσετε φυσικά δεν θα είναι, χρειάζεται να είναι πλήρης η απάντησή σας διότι θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε ελάχιστα λεπτά δεν τολμώ να σας πω ένα ο καθένας η κυρία Ριέρα Μαντουρέλ πρώτη, μετά η κυρία Καλβάλιο και μετά ο κύριο Σκίνερ. Τερέζα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω κυρίως ε, τον κύριο Σμιθ για την παρουσία του εδώ. Πολλά από τα θέματα που ανέφερε τα γνωρίζουμε και θα είναι λόγος και αφορμή συζήτησης όλον αυτό το χρόνο που θα έχουμε μπροστά μας, ενώπιόν μας. Και όχι μόνο θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε που για τις κοινωνικές επιστήμες και για την ασφάλεια που πρέπει να παραμείνουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο είναι ένα θέμα επί του οποίου υπάρχει γενικότερη συνένεση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και όλοι οι υπαΐοντες θα πρέπει να δρούμε σε αυτό το ενωμένο ενιαίο πλαίσιο και οι κοινωνικές επιστήμες αφορούν την ασφάλεια αλλά αφορούν και όλες τις άλλες και οποιασδήποτε άλλες προκλήσεις που εμπεριέχονται και υπάγονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και έτσι πιστεύουμε ότι και η έρευνα για τις κοινωνικές ε, επιστήμες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες μπορούν να έχουν μια ξεχωριστή βάση. Είναι ευκταίο λοιπόν και θετικό για όλη τη δομή του προγράμματος πλαισίου να ξεχωρίζουμε αυτά τα θέματα και αυτά τα πράγματα που όπως την κοινωνία και την ε, δυνατότητα αριστείας και υπεροχής ε, από τα κράτη-μέλη όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης που είναι γενικόλογη και ένα αμίγμα όχι τόσο εξειδικευμένο και που φαίνεται ένα μείγμα χίδιν όπου σε έναν ασκό έχουν ρηχθεί πολλά τέτοια στοιχεία και που εδώ πρέπει να δούμε και τον εγκάρσιο χαρακτήρα τους και έχουν επίπτωση σε όλο το πρόγραμμα πλαίσιο. Είναι πολύ πιο σαφής λοιπόν η πρόταση που γίνεται από τις εκθέσεις μας και που συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη με την κυρία Καρβάλιο και εν πάση περιπτώσει οπωσδήποτε θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε όλα αυτά και έτσι αυτό θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Grazie a lei, e a te, eh, e Λοιπόν, η κυρία Καρβάλιο θέλει μια σύντομη παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την ε, ε Κομισιόν του Γενικού Εθνητή Ρόμπερτ Σμίθ για τα σχόλιά του. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές όλοι ε, θέλουμε να πάμε προς την ίδια κατεύθυνση έτσι ώστε να αποκτήσουμε ένα απλό, ευέλικτο, καλά χρηματοδοτημένο ε, πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία. Τα μόνα σημεία ε, διαφωνίας, τα ανέφερε ήδη προλελήσα σας συνάδελφος Μαδουρέλ, αφορά την κοινωνική πρόκληση 6, καθώς επίσης και την, την απέτηση συμμετοχής, αν θα είναι πρώτος πυλώνας ή αν θα γίνει ε, στο, αν θα πάει στον υπαριθμό 6 όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν πάση περιπτώσει θα έχουμε περαιτέρω συζητήσεις για το θέμα αυτό κατά τα λοιπά πιστεύω ότι είμαστε ευθυγραμμισμένοι με το Συμβούλιο και την Κομισιόν τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι το εξής Αυτό το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά φιλόδοξο. Και στο Κοινοβούλιο έχουμε ε, επίσης προσθέσει και άλλες φιλοδοξίες. Ε, δηλαδή πολλά στοιχεία στα ήδη πολλά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να μπορέσουμε να είμαστε επιτυχείς όσον αφορά τον ορίζοντα 2020 θα θέλουμε, χρειαζόμαστε απαραίτητη, την, την απαραίτητη χρηματοδότηση. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θα αγωνιστούν έτσι ώστε ο Ρίζων 2020 να έχει την απαραίτητη χρηματοδότηση και ευελπιστούμε ότι θα επιτύχουμε συμφωνία όσον αφορά ε, χρηματοδότηση που θα είναι στο ύψος ε, των περιστάσεων και των φιλοδοξιών. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο ε, σύμφωνο και επομένως από τη στιγμή που όλοι συμφωνούμε ότι είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σημαντικό. Θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε έτσι ώστε η χρηματοδότηση να είναι σωστή. Ο Πίτερ Σκίνερ, τελευταία παρέμβαση. Σχετικά με αυτά τα οποία ανέφερα προηγουμένως δεν ε, μπόρεσα να απαντήσω. Κύριε Βιδάλ Κουάδρας, αναφέρατε ε, την βασική έρευνα και είπε ότι είναι απαραίτητη. Συμφωνώ μαζί του. Αυτό που λέω εγώ όμως είναι ότι δεν θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα μονάχα ε, σε θέματα όπως είναι τα ε, Marie Curie και όλα τα χρήματα τελικά να μπαίνουν, ε, να πηγαίνουν στην βασική έρευνα η οποία δεν μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα της καινοτομίας που θα πρέπει να είναι κοντά στην αγορά. Το θέμα είναι το πώς παίρνει την επιστήμη, πώς την εφαρμόζεις έτσι ώστε η οικονομία να ωφεληθεί ε, έτσι ώστε να ωφεληθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το σημαντικό. Και επομένως αντί να βάζουμε όλα τα χρήματα σε παραδοσιακές περιοχές έρευνας ε, θα πρέπει να ε, δώσουμε τα χρήματα με σωστό τρόπο γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολλά η ιδέα της ε, προσέλκυσης ε, ιδιωτικών ε, χρηματοδοτήσεων ήταν έτσι ώστε να υπάρχει μια δυνατότητα εξισορρόπητης αλλά τα venture τα capitals και τα κεφάλαια κινδύνου βεβαίως είναι πιο δύσκολο να, να, τα διαχειριστεί κανείς. Οπωσδήποτε όλα αυτά όμως θα πρέπει να αναφέρονται σε αυτή τη δέσμη και βεβαίως θα πρέπει και προκύπτει σαφώς ότι δεν αρκεί η βασική έρευνα. Πρέπει να είμαστε πιο κοντά στην ε, αγορά ε, και κατά αυτήν την έννοια θα πρέπει να δούμε ε, και την πυρηνική φυσική και την χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Αλλά και εκεί χρειάζεται βεβαίως βασική έρευνα και εκεί και με το σκεπτικό αυτό οδηγούμαστε στην ενεργειακή αυτάρκεια που είναι ένα θέμα το οποίο όλους μας απασχολεί αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σμιθ ε, θέλει να, ε, να πάρει το λόγο. Του δίνουμε τη δυνατότητα να απαντήσει, γιατί βεβαίως θέλουμε να δουλέψουμε μαζί ε, προς την ίδια κατεύθυνση η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και επομένως και τον ευχαριστούμε κιόλας που είναι τόσο στη διάθεσή μας. Θα είμαι πολύ σύντομο. Ξέχασα απλώ να απαντήσω στο θέμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογία και Καινοτομία. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις που άκουσα από τους κυρίους Λαμπέρ και Γιώχανσον ότι το ανακαλύπτεται σιγά σιγά αυτό το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Γενοτομίας και είναι μια ενδιαφέρουσα και πολλά υποσχόμενη ιδέα για να έχουμε αυτό το τρίπτυχο της γνώσης. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα λοιπόν η προσοχή που δίνεται σε αυτό το Ινστιτούτο διότι θα είναι ένα εργαλείο εντός του ορίζοντα 2020 το οποίο θα συνεισφέρει στην καινοτομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Λοιπόν, συμπληρώνεται η συζήτηση για όλη αυτή τη δέσμη μέτρων και ευχαριστώ και τον κύριο Τσίτσεστερ, ο οποίος προείδρευσε για το μισό της συνεδρίασης. Αυτή λοιπόν η μακρά συζήτηση ολοκληρώνεται με τις προθεσμίες κατάθεσης τροπολογιών, που είναι διαφοροποιημένες για τις εκθέσεις Ρέιρο Μαντιλάρ και Σκίνελ, 3η 26 Ιουνίου 12 το μεσημέρι. Εκθέσει Έλερ και Λάμπερτ. Τετάρτη 27 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι. Και για τις εκθέσεις Καρβάγιο και Ματίας, 5η 28 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι. Η συζήτηση στη συνέχεια θα γίνει για εξέταση τροπολογιών σε δύο συνεδριάσεις. Πρώτη εξέταση των τροπολογιών Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου. Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους ε, συμμετείχαν, σκιώδεις, εισηγητές και ομιλητές και να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση εδώ. Το δεύτερο τμήμα αφορά μια άλλη δεσμή μέτρων, η οποία μπορεί να μην ε, συμπεριλαμβάνεται στον ορίζοντα 2020, αλλά σίγουρα συνδέεται. Είναι το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για το 2014-2020, το COSME. Το ρόλο έχει ο εισηγητής, ο κύριος Κρόιτσμαν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για το μόνο ειδικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μετά από την μετάθεση κέντρου βάρους για την καινοτομία όσον αφορά τον ορίζοντα 2020 έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ για τη συνεργασία την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο σχέδιο έκθεσής μου κάνω μια σειρά προτάσεων ώστε αυτό το σχέδιο να μπορέσει να γίνει πιο εξειδικευμένο. 2,5 δις ευρώ είναι τα κονδύλια αυτού του προγράμματος, σχετικά περιορισμένα, αν δει κανείς όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το τοπίο τους. Γι' αυτό προτείνω σε τρεις άξονες να επικεντρωθούμε για τους οποίους η δική μου ομάδα καταβάλει προσπάθειες εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Μείωση του γραφειοκρατικού βάρους, προσπελασιμότητα στη χρηματοδότηση, διευκόλυνση της προσπελασιμότητας της πρόσβασης στις αγορές. Προτείνω για τη μείωση γραφειοκρατικού βάρους η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα φιλόδοξο ε, στόχο για την ε, ε, ανακούφιση και να υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης αυτού του εγχειρήματος σε διαφοροποίηση με την τελευταία μας ε, ε, στοχοθέτηση αυτό σημαίνει και με νέα νομοθεσία θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη η γραφειοκρατική επιβάρυνση που παρόλα αυτά πρέπει να επιτυγχάνεται από κοινού στις ε, ενώσεις και συλλόγους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει ποιοτικοί στόχοι να εντάσσονται. Σε συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ποσοστοποιήσουμε τους στόχους. Δεν είναι χωρίς πρόβλημα αυτό. Και το πόσο μπορούμε να το καταφέρουμε. Το θέμα όμως είναι οι ποιοτικοί στόχοι να καθοριστούν ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει από κοινού να προβληματιστούμε πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Επιπρόσθετα μπορεί να αποφευθεί η, γραφειοκρατη... η γραφειοκρατία όταν μέσω των μελετών επιπτώσεων συστηματικά εφαρμόζουμε τα στοιχεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βλέπουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις τέτοιων ρυθμίσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεων. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα μέσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δεύτερη δυνατότητα, προσπελασιμότητα σε χρηματοδότηση. Εδώ μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά το πρόγραμμα, ώστε να καλυφθούν τα κενά και ε, οι ελλείψεις ε, που υπάρχουν στην αγορά. Χρήση κεφαλαιοκρατικών, κεφαλαιακών ε, μέσων και εργαλείων μέσω του Innovation Program που έχει δείξει ότι ήταν πραγματικά καλό. Έχουν μοχλευτική επίπτωση και είναι πολύ καλά αυτά τα προγράμματα και μέτρα για την δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης. Η πείρα έδειξε ότι η ζήτηση για αυτά τα μέσα και εργαλεία κατά κανόνα υπερβαίνει κατά πολύ τα πλαίσια του προγράμματος. Προτείνω 55,5% ε, να καλύπτεται από αυτό το πρόγραμμα για τα χρηματοδοτικά μέσα που θα προβλέπονται. Στην περίπτωση που, αν δεν, που δεν αντληθεί αυτός ο όγκος, τότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να παρέμβει. Ωστόσο ανησυχώ κάπως για τον κατακαιρματισμό των χρηματοδοτικών μέσων για τον ορίζοντα 2020 που ε, αυξάνει την περιπλοκότητα για όσους εμπλέκονται. Είναι σημαντικό να υπάρξουν διαχωριστικές γραμμές και διαφοροποιήσεις και από την άλλη πλευρά μέσω επαφών να βοηθούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρουν τους συνδέσμους τους και τους εταίρους τους. Είναι σημαντικό το εγχείρημα για την καινοτομία, διότι η οικονομία μέσω της ε, ε, δυνατότητας ε, να μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές δεν θα πρέπει να ε, οι προσπάθειές τους να αποβαίνουν άκαρπες. Το πρόβλημα αυτό για 150.000 ευρώ για τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Κατά τα άλλα αντανακλά αυτό και τον συμβιβασμό που πιστεύουμε ότι ε, σε σχέση με το Συμβούλιο επιτυγχάνεται. Τρίτον, θα πρέπει να συνεισφέρει το πρόγραμμα αυτό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην ενιαία εσωτερική αγορά και στις αγορές γενικότερα. Η επιχειρηματικότητα και η διαδικτύωση είναι σημαντική. Το δίκτυο αυτό με το πρόγραμμα SIP εισήχθη και έχει αναπτυχθεί περαιτέρω από τότε που δημιουργήθηκε. Όμως το δίκτυο αυτό δεν έχει επιτυχία, η ίδια και ίση επιτυχία σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δούμε το δίκτυο αυτό που πρέπει να έχει καλύτερη κάλυψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει τις διαφορετικές δομές και υποδομές στα κράτη-μέλη και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση αυτής της δικτύωσης. Συγκεκριμένα ε, μέτρα ε, που μπορούν να βοηθήσουν πρέπει να υποστηριχθούν εφόσον ε, ε, δεν επιβαρύνονται οι υπηρεσίες στα κράτη-μέλη ή δεν υπάρχουν επικαλύψεις. Επίσης, ε, σε σχέση και με τις παραγγελίες, η τυποποίηση είναι σημαντική πριν από τη λήψη τέτοιων μέτρων πρέπει να προβεί σε μελέτη των υφιστάμενων μέτρων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μελέτη επιπτώσεων. Αυτή η ανάλυση θα πρέπει να γίνει μέσα στο πλαίσιο του ΣΥΠ, προγράμματος ΣΥΠ και να ολοκληρωθεί εκεί. Συνιστάται λοιπόν να υπάρξει συνέχιση αυτής της προσπάθειας, συνέχεια αυτής της προσπάθειας. Παράλληλα με αυτές τις προτεραιότητες έχω στην έκθεσή μου πέντε γενικούς στόχους το πρόγραμμα θα πρέπει να στρέφεται προς όλες τις μικρομεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει όχι μόνο διασυνοριακά να περιορίζεται σε αυτές τις επιχειρήσεις που δρούν διαμεθοριακά, υπάρχουν σημαντικά κριτήρια η παραγωγή πρόσθετης ευρωπαϊκής αξίας. Αλλά αυτή η πρόσθετη ευρωπαϊκή αξία μπορεί να υφίσταται στην αντιστάθμιση ελλείψεων στο τοπικό περιφερειακό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών και μέτρων. Θα πρέπει διατομεακά να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες που το δυνατόν θα έχουν ωφέλη, θα, θα οδηγούν σε ωφέλη το δυνατόν σε περισσότερες ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να υπάρχει εδώ η παραγωγή ευρωπαϊκής πρόσθετης αξίας Ωστόσο, είναι σημαντικό ο τουρισμός να δούμε ότι στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να ε, ξεχωρίζεται. Το κόσμο δεν είναι τουριστικό πρόγραμμα. Ξέρω, δεν έχουμε πρόβλημα, Επίτροπε, αν ε, το δυνατόν περισσότερες αιτήσει ε, υποβάλλονται και το δυνατόν περισσότερες ιδέες στον τομέα του τουρισμού προωθούνται. Αυτό είναι κάτι το αυτονόητο και πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και να προωθείτε. Δεν ξέρω όμως αν τομεακά μία τομεακή ε, επιλογή πρέπει να γίνεται. Ξέρω ότι υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις και σε άλλους τομείς. Θα ε, οδηγούσε κανείς, ε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα υπήρχαν παρεμβάσεις που θα αμφισβητούσαν μία και μόνο τομεακή επιλογή. Γι' αυτό θα πρέπει καλύτερα να δούμε τους επιμέρους τομείς σε εξειδικευμένα μέτρα που θα πρέπει να ε, λαμβάνονται και αυτό κάνω στις τροπολογίες μου. Οι ενώσεις και σύλλογοι μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να εντάσσονται με καλύτερο τρόπο σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Με καλύτερη ε, διαμόρφωση κόστους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έτσι να υπάρχει συμβουλευτική δραστηριότητα για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας γνωρίζω ότι υπάρχουν επιφυλάξεις σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτές τις προτάσεις. Είμαι πρόθυμος από κοινού με τους κοιόδης εισηγητές να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε πώς η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να διασφαλιστεί χωρίς να υπάρχει περιττή επιβάρυνση που θα προκαλείται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποφασίζει βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μπορεί να έχει νόημα να υπάρχουν προτάσεις και κίνητρα που θα υποβάλλονται από τις ενώσεις και συλλόγους μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό θα ήταν θετικό και έτσι θα πρέπει να λαμβάνονται αυτά υπόψη. Τέταρτον, το πρόγραμμα δεν θα πρέπει μόνο να περιορίζεται στη φάση ανάπτυξης, αλλά να συμπεριλαμβάνει στον κύκλο ζωής όλες τις φάσεις ενός κύκλου ζωής. Ιδιαίτερα η ίδρυση, η μεταφορά, μετάθεση νέων ε, δυνατοτήτων κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις απειλούνται στην Ευρώπη επειδή δεν υπάρχουν ε, ε, διάδοχες ε, καταστάσεις που να διασφαλίζουν επενδύσεις σε αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι όμως σημαντικό να δούμε τη διασφάλιση της ευημερία μέσω της διασφάλισης των επενδύσεων και της συνέχειας της επιχειρηματικής δράσης. Ολοκληρώνω άμεσα Πρόεδρε και έχουμε φιλόδοξους στόχους και είναι σημαντικό λοιπόν να ληφθούν αυτοί υπόψη και να σκεφτούμε κατά πόσον αυτό το πρόγραμμα μπορεί να λάβει υπόψη αυτές τις συνιστώσεις. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ξέρετε, όταν φτάνουμε στο τελευταίο σημείο, μετά δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Λοιπόν, ε, σκιώδης του, του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Γιώργαν Κρότσμαν για τη σκληρή δουλειά που έκανε όσον αφορά την προσέγγιση για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι η πρόταση είναι πολύ καλή ε, και θα είναι καλή και ευεργετική για όλες τις ευρωπαϊκές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα COSME εστιάζεται στην μείωση του διοικητικού ε, άχθους και βελτιώνει την πρόσβαση στην αγορά για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο αυτές οι οποίες έχουν διασυνοριακές συναλλαγές ή αυτές που ασχολούνται με τον τουρισμό όπως στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Ε, η μείωση του διοικητικού κόστους είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουμε την προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας που αποτελεί ένα κυρίο πρόσκομα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, το κατόφλι για, ε, για τα εγγυημένα δάνεια ε, και για την επιλεξιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ορίζοντα 2020 θα καλυφθούν από το κόσμο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, βλέπω με ευχαρίστηση ότι ε, έχει καλά στοιχεία όλη αυτή ε, η προσπάθεια. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα από τα κυρίαρχα σημεία τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουμε, δηλαδή τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της, δικές τους, της δικιάς τους χώρας. Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία σε όλες τις χώρες. Ε, θα πρέπει ε, επίσης ε, όλοι οι πόροι που είναι απαραίτητοι να χρησιμοποιηθούν ο προϋπολογισμός δυστυχώς ο οποίος έχει δοθεί δεν αποδίδει την πολιτική βαρύτητα του θέματος. Το κόσμο, όπως είπε και ο κύριος Κρόσμε, έχει προϋπολογισμό 2,5 ε, δηλαδή 0,5% ε, ε, των, του πολιετού του δημοσιονομικού πλαισίου. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και αν θέλουμε πραγματικά να πούμε και αν πιστεύουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το όχημα για την άδειξη της Ευρώπης, θα πρέπει οπωσδήποτε να φτάσουμε από το 0,5% στο 2,5% του προπολογισμού. η πρόσβαση ή μάλλον η αδυναμία πρόσβαση στην ε, ε, τραπεζική πίστη και στα χρηματοπιστωτικά ε, ιδρύματα είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω και εγώ μια παρέμβαση ως και όδηση για το θέμα αυτό. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κρόιτσμαντ για τα όσα έκανε. Πραγματικά πολύ αναλυτική δουλειά, πολύ εύστοχη. Λαμβάνει υπόψη της και όλα τα προβλήματα του τομέα και για τις ακροάσεις που διοργάνωσε και το προσκευαστικό του έργο. Όπω έλεγε και ο συνάδελφος του ΕΛΚ, θεωρώ και εγώ ότι δεν υπάρχει σχέση μετά ξύ αρκετών δηλώσεων που κάνουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσει και αυτό το 0,2% των πολιετών δημοσιονομικών προεπτικών που ε, είναι για το κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο. Επίσης θεωρώ ότι όπως ακούστηκε ε, και σε κάποιες συζητήσεις που κάναμε στο Στρασβούργο, Εάν η κάθε μικρομεσαία επιχείρηση προσλάμβανε έναν επιπλέον εργαζόμενο ή εργαζόμενη, θα είχαμε εν μέρη λύσει το πρόβλημα τη ανεργία τη Ευρώπη. Αναφερόμαστε λοιπόν σε ένα τομέα ο οποίο πράγματι μπορεί να απορροφήσει και ε, σε μικρέ ίσω ποσότητε, αλλά πλασιαζόμενε με τον αριθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γίνονται μεγάλε, ε, πολύ μεγάλο αριθμό ανέργων. Γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι το τμήμα του κόσμου, των πόρων του κόσμου που δίνονται από τα χρηματοδοτικά μέσα είναι ελάχιστο και ίσως θα έπρεπε να επανεξετάσουμε αυτή την κατανομή εντός του προγράμματος. Οι άλλες δράσεις είναι σημαντικές, κατάρτιση, ε, και όλες οι παράπλευρες δράσεις αν θέλετε, αλλά δεν θα πρέπει να αφαιρούμε πόρους από το βασικό ε, έργο, από τα χρηματοδοτικά μέσα και νομίζω ότι θα το πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το ζήτημα. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα το οποίο ήδη προέκυψε στη συζήτηση ε, σήμερα, σε αυτά τα λίγα λεπτά που συζητήσαμε, και αφορά τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε και δράσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό το διεθνές στοιχείο, όχι μόνο για τις μεγάλες, αλλά και για τις μικρές και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που μπορούν να διαστηριοποιηθούν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα προϊόντα τους και αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης σημαντικό είναι να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση για τα χρηματοδοτικό μας προγράμματα. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί και σε εσά, αλλά εμβαθύνοντας αυτό το πρόγραμμα με κάποιους ε, ενδιαφερομένους ε, του τομέα των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διαπίστωσα ότι πολύ συχνά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία είναι οι διαμεσολευητές ανάμεσα στα προγράμματά μας ε, και ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή στο ταμείο που τους χρηματοδοτεί, δεν ε, δίνουν αυτές τις πληροφορίες στους ενδιαφερομένους, διότι ενδιάμεσα βρίσκεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο δεν ενδιαφέρεται να χρηματοδοτήσει αυτά τα μέσα και εργάζεται με μεγαλύτερη ευκολία και ίσως με μεγαλύτερο κέντρο, κέρδο συγγνώμη, με άλλα μέσα. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δημοσιοποιήσουμε τα προγράμματα αυτά, ακόμα και αν δίνουν λίγου πόρους. Επομένως θα πρέπει να υπάρξει κάποια τροπολογία και του και εγώ θα πρέπει, ε, θα ήθελα να πάμε προ αυτή την κατάσταση. Και θεωρώ επίσης ότι τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και να είναι και ισχυρά, διότι αλλιώς δεν φτάνουν ε, στους ενδιαφερομένους. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιμένουν, οι τράπεζες δεν ενδιαφέρονται να τα γνωστοποιήσουν, να τα δημοσιοποιήσουν και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα αποφύγουμε. Δεν συμφωνώ σε όλα με τον εισηγητή για το θέμα του τουρισμού. Θεωρώ ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι στερούμε πόρους από κάποιους. Κάποια τουριστικά προγράμματα είναι διατομεακά, διότι υπάρχει ο τουρισμός και επιχειρήσεις που συνδέονται με τον κόσμο του τουρισμού. Θα πρέπει λίγο να δούμε την Ευρώπη ε, σε όλη τη την ποικιλομορφία και θεωρώ ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε λίγο και αυτή την ψυχή. Και μια τελευταία μου παρατήρηση για αυτό το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων, το European Enterprise Network, στο οποίο ε, είναι κάτι ε, για το οποίο θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει λίγο πιο ε, συνεκτική δουλειά. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες. Εάν θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτό το δίκτυο και με πόρους, θα πρέπει να κατανοήσουμε πώς είναι φτιαγμένο αυτό το δίκτυο και πώς λειτουργεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τον εισηγητή για τη δουλειά του, διότι μας διευκολύνει και εμάς ως σκιώδης εισηγητής, διότι πολλά τα όσα θέλουμε να πούμε τα έχει πει στο κείμενό του. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, ούτε εγώ δεν σεβάστηκα το χρόνο και ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Βινταλ Κουάντρας. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, είναι πάνω από 90% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα μεταξύ τους. Δυσκολίες για να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές, γραφειοκρατική επιβάρυνση που είναι όλο και μεγαλύτερη και επιδεινώνει τα πράγματα. Για όλα αυτά είναι σημαντικό ένα πρόγραμμα να στοχεύει σε αυτό τον τομέα που να είναι το δυνατόν πιο αποτελεσματικό. Το σχέδιο έκθεσης που μόλις ο συνάδελφος Κρόισμαν παρουσίασε περιέχει μια σειρά βελτιώσεων που χωρίς αμφιβολία είναι σωστές για παράδειγμα η εισαγωγή συγκεκριμένων αναφορών στην Small Business Act που πρέπει να είναι τα ορόσημά μας για την ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άλλο παράδειγμα που πρέπει να τονίσουμε είναι οι τροπολογίες που στοχεύουν στο να βελτιώσουν το δίκτυο των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, Enterprise Europe Network, αποτελεσματική δικτύωση και δίκτυο, αλλά πρέπει και αυτό να βελτιωθεί και να ενδυναμωθεί ο ρόλος που έχουν οι οργανώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λόγω του μεγέθους τους πρέπει να μπορούν να δρουν από κοινού και δικτυωμένες σε οι οργανώσεις αυτές πρέπει να μπορούν να ε, αποτελέσουν δυνατότητα εκμετάλλευσης και ενδυνάμωσης ιδιαίτερα σε εκείνους τους τομείς όπου συνεισφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημαντικά για την δημιουργία του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και στον τουριστικό προφανώς τομέα επίσης προφανώς και εγώ ίδιος ε, συμφωνώ με την προσέγγιση και τη διαπίστωση ότι είναι ενδιαφέρουσες οι αναφορές στον τομέα του τουρισμού. Και αυτό επειδή είναι ένας από τους τομείς που πρέπει να εργαστούμε μέσα στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος αν θέλουμε να πετύχουμε αυτός ο κανονισμός σε μια περίοδο έκδηλης κρίσης στα κράτη-μέλη. Έχουμε ε, κράτη-μέλη με πάρα πολύ σημαντική παρουσία στον τουρισμό. Αν θέλουμε πραγματικά να συνεισφέρουμε στο να ενδυναμωθεί αυτή η συνιστόσα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το ευρωπαϊκό λοιπόν όραμα αυτό πρέπει έτσι να λειτουργήσει και έτσι να το προσεγγίσουμε. Μία συγκεκριμένη αναφορά στον τουρισμό είναι σωστή νομίζω σε αυτό το πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά το κατόφλι 150.000 ευρώ για δάνεια που θα μπορούν να εγγυώνται μέσω μέσων εγγύησης θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς σε αύξηση αυτού του κατοφλίου, μια και είναι χαμηλού επίπεδου. Και πρέπει να υπάρχει και σαφής δυνατότητα τα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν εθνικά ε, χρηματοοικονομικά μέτρα και ευρωπαϊκά στη διάθεσή τους. Ε, Ευχαριστώ. πολύ. Ε, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήδη σε γενικές γραμμές έγινε λόγος για σχεδόν όλα όσα εμπεριέχει αυτή η έκθεση. Η αλήθεια είναι σε γενικές γραμμές συμφωνούμε σε αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο εισηγητής για το θέμα της χρηματοδότησης. Η ανεπαρκής χρηματοδότηση ενός τόσο σημαντικού προγράμματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος της κινητήριας δύναμης στην Ευρώπη πρέπει να αυξηθεί. Πρέπει να αυξηθούν οι χρηματοοικονομικές δυνατότητες. Είναι αναγκαίο να κατανείμει τα κονδύλια έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με κάθε τομεακή δραστηριότητα για να ξέρουμε τι θα είναι και τι όχι στη διάθεσή τους. Και είναι αυτονόητο ότι πρέπει με θετικό τρόπο να μπορεί να αξιολογηθεί το θέμα της μείωσης της γραφειοκρατικής επιβάρηση όσον αφορά και την πρόσβαση σε ε, δυνατότητα να ενδυναμωθούν οι επιχειρήσεις και οι συνέργειες που πρέπει να υπάρχουν για την ε, ε, περιφερειακή και επαρχιακή κάλυψη των δράσεων αυτών των, επιχει... των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτό το χρηματοοικονομικό μέσο να μπορεί να χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση εγγυήσεων κεφαλαίου και για το κατόφλι του 150.000 ευρώ πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ χαμηλό για τις ανάγκες για τη χρηματοδότηση. Έγινε λοιπόν ε, μια συγκεκριμένη αναφορά για τον τουρισμό και πιστεύω ότι εισήγαγε με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια προσέγγιση υπό την έννοια ότι ο τουρισμός είναι, αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανταγωνιστικές και βιώσιμες που αποτελούν μέρος και τμήμα της δημιουργίας του ΑΕΠ σε κάθε χώρα με εκπληκτικό τρόπο πιστεύει κανείς ότι μόνο στις χώρες του Νότου ή στις ε, καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες μπορούν να λειτουργήσουν. Αν δούμε όμως πώς συνδιαμορφώνουν το ΑΕΠ σε κάθε χώρα θα μπορούσαμε να εκπλαγούμε. Ιδιαίτερα ο τουρισμός λοιπόν πάλι αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανταγωνιστικές που πρέπει να ε, διασφαλίζουν την αηφορία τους και τη βιωσιμότητά τους. Δημιουργούν απασχόληση αυτές οι επιχειρήσεις και ανταποκρίνονται στις ιδιομορφίες και ανάγκες της κοινωνίας για τον τουρισμό και τις συγκεκριμένες αυτές ε, δραστηριότητες. Θα υποβάλουμε, θα καταθέσουμε συγκεκριμένες τροπολογίες που θα στοχεύουν στο να βελτιωθεί η έκθεση που παρουσιάζει ο εισηγητής και πιστεύουμε ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να δώσουμε από πλευράς κονδυλίων ε, τα αναγκαία κονδύλια ώστε το πρόγραμμα αυτό να ανταποκρίνεται ε, στη σπουδαιότητά του και στις ανάγκες του. Διαφορετικά δεν θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Ο κύριος Χέρμπερ νομίζω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο λεπτά σας δίνω μονάχα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή κύριο Κρότσμαν καθώς επίσης και τα υπόλοιπα μέλη της, Ευρωπη... της Επιτροπής σας ε, για την στήριξη που έδωσαν στο πρόγραμμα COSME στο σχέδιο έκθεσης του ο κύριος Κρότσμαν αναγνωρίζει την ανάγκη στήριξης των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως δε την πρόσβαση στην αγορά, στη χρηματοδότηση και τη μείωση της, ε, του διοικητικού άχθους ε, για όλες τις επιχειρήσεις γενικά τώρα. Προτείνει ο εισηγητής να απλουστευτούν περαιτέρω διαδικασίες μέσω απαρίθμησης των στοιχείων. Βεβαίως αυτό είναι χρήσιμο, αλλά πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο θα διατηρηθεί μέχρι το 2020. Γι' αυτό δεν θέλουμε να δυναμητήσουμε την απαραίτητη ευελιξία του προγράμματος COSME και σας υπενθυμίζω ότι το πρόγραμμα SIP ε, ακριβώς ε, ε, θεωρήθηκε πολύ καλό όσον αφορά την ευελιξία του για την πρόσβαση στην αγορά οι προτεραιότητε που αναφέρει ο κ. Κρότσμαν βρίσκουν θετικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω θα πρέπει να υπογραμμιστεί η προστιθέμενη αξία καθώς επίσης ε, και το ο αντίκτυπος, ε, ο που θα πρέπει να έχουν οι δράσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, βεβαίως από τη στιγμή που όλε, όλα τα θεσμικά όργανα θα εγκρίνουν την πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορέσει το πρόγραμμα αυτό το οποίο είναι φιλόδοξο να δώσει ε, αποτελέσματα. Ε, εμείς θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη ε, σημασία και βάρος στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Η ποιοτική διάσταση, η διαρκής ποιοτική υπογράμμιση μας ενδιαφέρει περισσότερο. Δύο παρατηρήσεις επίσης. Ε, είναι γεγονός ότι για δάνεια πάνω από 150.000 ευρώ ε, το σύνολο των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα αφορά η πρόταση οπωσδήποτε μειώνεται αλλά θα πρέπει να το ξαναδούμε. Με το παρόν χρηματοδοτικό πλαίσιο μας ενδιαφέρει να ε, είμαστε σύμφωνοι με τις αρχές ε, της ε, ανταγωνιστικότητας. Πρόσβαση στην αγορά, το είπατε κι εσείς, είναι προτεραιότητα. Πιστεύουμε ότι το δίκτυο, το Enterprise Network μπορεί να παίξει ρόλο, αλλά βεβαίως μπορεί περαιτέρω να βελτιωθεί. Συμφωνούμε μαζί σας. Είναι κάτι το οποίο διαρκώς θα πρέπει να, να βελτιώνεται. Έχουμε πάντως και τους εταίρους που απαντούν εθελοντικά στις ε, εκκλήσεις που κάνουμε στην αγορά, αλλά καταλάβαμε τι θέλετε να πείτε. Τέλος, πολύ σύντομα, χαιρόμαστε για την αναφορά που κάνετε στο ESBA Επίσης, χαιρόμαστε για την αναφορά που κάνετε στις ειδικέ δραστηριότητες σε περιφέρειες με πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά λαμβάνοντας την αναφορά στις συνθήκη της Λισαβόνας και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι διαφορετικός ε, στόχος από τη βιομηχανία, πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να γίνει ειδική αναφορά στον τουρισμό. Τέλος, η διαβούλευση με, τον επιχειρήσεων, με τις επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμφωνούμε απολύτως μαζί σας. Το κάνουμε ήδη. Κάθε δύο μήνες οργανώνουμε ε, συναντήσεις ε, με τους εκπροσώπου εκπροσώπους ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μία φορά το χρόνο έχουμε συνέλευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα κάνουμε όλα αυτά ε, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε να λύσουμε χωρίς υπερβάλλουσα γραφειοκρατία όλα τα θέματα τα οποία συνδέονται με, την, ε, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την την ανταγωνιστικότητά τους, συγγνώμη, την αντιπροσωπευτικότητά του κλπ. Και εδώ μην ξεχνάμε ότι το καλύτερο είναι ο εχθρό του καλού. Ε, Βεβαίω ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ε, δύσκολε επιλογέ. Ξέρετε την πρόταση τη Επιτροπή. Καταλάβαμε όμω και εμεί αυτό που θέλατε να πείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη που μα δίνετε σε αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Κρόιτσμαν τώρα. σα παρακαλώ να είστε σύντομο, γιατί έχουμε ένα ακόμα σημείο στην ημερήσια διάταξη και αν ε, είναι δυνατόν. Θα ήθελα να δώσουμε και τη δυνατότητα στον κύριο Κάλφιν να παρουσιάσει την έκθεσή του, γιατί αύριο έχει μια πολύ σημαντική συνεδρίαση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλήστιο. Παρακαλώ. Να ευχαριστήσω για τι θετικέ ε, τοποθετήσει. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη ότι τόλμησα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σκεφτούμε για τον ίδιο τομέα. Έχουμε ήδη μέσα εντός αυτές τις προτάσεις, δεν είναι εκτός. Όμως το πρόβλημα είναι αν ονομαστεί, προσδιοριστεί ένας τομέας μόνο και άλλοι θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Δεν έχω καμία αντίρρηση να προαθεί ο τουρισμός. Το κατανοώ αυτό ότι πρέπει να γίνει. Δεν ήταν κάτι το οποίο διαφωνούσα εγώ, αλλά έχει νόημα, πρέπει να δούμε να γίνεται κάτι τέτοιο. Εν πάση περίπτωση δεν υπάρχει πρόβλημα. Να πω δύο λόγια για τον προπολογισμό. Και Άλλοι ανέφεραν το 15% είναι πολύ λίγο ως ποσοστό για τον ορίζοντα 2020. Το 20% δεν είναι δεσμευτικό. Το ερώτημα που τίθεται και που πρέπει όλοι να προβληματιστούμε από αυτού είναι δεν θα είχε νόημα αντί 15% να κάνουμε λόγο για 8,5 δις ή όπως θέλει το Συμβούλιο ίσως για να το αυξήσουμε σε 20 και να πούμε το κόσμο να είναι 5 δισεκατομμυρίων από το 0,2% στο 0,5% και αυτό ουσιαστικό θα ήταν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να αυξήσουμε και το κονδύλιο για αυτές. Θα έχουμε περισσότερα κονδύλια διαθέσιμα. Είναι σαφές λοιπόν. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς κάποιες δεσμευτικές αναφορές. Αλλά προτού αρχίσουμε να αναφέρουμε κάποιες μη δεσμευτικές στοχοθετήσεις στον ορίζοντα 2020 σκόπιμο θα ήταν να προβληματιστούμε από κοινού τι πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ για τα θετικά λόγια από όλους όσους ε, έλαβαν τον λόγο. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστούμε. Τροπολογίες 12 ε, το μεσημέρι 20 Ιουνίου. Θα θέλαμε τώρα να δώσουμε τον λόγο στον συνάδελφο Κάρινς ε, για να μας πει ε, ποιες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά το μηχανισμό ανταλλαγής ε, πληροφοριών κλπ. για τις διακυβερνητικές συμφωνίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φαντάζομαι ότι όλοι θυμούνται ότι στην Επιτροπή μας εγκρίναμε όσον αφορά τον μηχανισμό ανταλλαγής ε, πληροφοριών ε, σχετικά με τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών Μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας πολύ ε, συγκεκριμένα μέτρα στα οποία κυριαρχούσε η διαφάνεια στον τομέα της ενέργειας πρέπει να δούμε εάν οι επιχειρήσεις ευθυγραμμίζονται με την πολιτική ενέργειας. Κυρίως όταν αναφερόμαστε σε πρόσβαση τρίτων χωρών στην υπο στις υποδομές ενέργειας. Υπήρξαν τριμερείς διάλογοι. Όμως, παρά την απόφαση του προηγούμενου Φεβρουαρίου του Συμβουλίου, βάσει ε, η συντηρητική πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου φαίνεται ότι εξακολουθούν να λένε δεν θέλουν αυτήν την νομοθεσία με οποιαδήποτε μορφή. Ε, είπαν ότι η πρόταση ε, που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την οποία ενίσχυσε το Κοινοβούλιο δεν τη θέλουν φαίνεται στο Συμβούλιο. Λοιπόν, κατάφερα να επιτύχω ένα συμβιβαστικό κείμενο. Συμβιβαστικό κείμενο το οποίο βεβαίως δεν ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Επιτροπής μας, αλλά είναι καλύτερο από το τίποτα. Ε, δεν ανταποκρίνεται κυρίως όσον αφορά τον έλεγχο ε, συμμόρφωσης εξάντε. Η Κομισιόν ε, είπε ότι θα κοιτάξει λίγο τα στοιχεία αυτά πριν υπογράψει. Το Συμβούλιο όμως δεν συμφώνησε καθόλου. Δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο στην ε, νομοθεσία. Εν πάση περιπτώσει εμείς ε, βρήκαμε κάποια στοιχεία τα οποία προωθούν λίγο το θέμα. Έχει μπει και μία ρήτρα αναθεώρησης έτσι ώστε σε τρία χρόνια να δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Είναι δύσκολη λοιπόν η κατάσταση το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν φαίνεται ότι δεν μπορούν να συμφωνήσουν απέναντι στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δηλαδή δεν μπορεί να συμφωνήσει. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα συμβαστικό κείμενο και προτείνω λοιπόν εμείς ως πλευρά Κοινοβουλίου να πάμε σε συμφωνία πρώτης ανάγνωσης γιατί τελικά το ερώτημα είναι το εξής. Ε, δεν είναι καλύτερα κάποια μορφής νομοθεσία παρά καμία μορφής νομοθεσία. Ε, εάν έχουμε κάποια νομοθεσία σαν βάση μπορούμε σιγά σιγά και εν το χρόνο να την τροποποιήσουμε. Αν δεν έχουμε τίποτα δεν θα μπορέσουμε. Θα ξεκινάμε πάντα από το μηδέν. Ε, προτείνω λοιπόν ότι είναι εδώ το μη χείρον βέλτιστον. Να ευχαριστήσω τους αδέλφους που συμμετείχαν στον τριμερή διάλογο, στο τελευταίο τριμερή διάλογο ε, μετά από δικιά μου επιμονή καταφέραμε να δούμε κάποια στοιχεία και ο πρόεδρος μάλιστα ήταν τόσο αγχωμένος και τόσο πολύ δεν ήθελε να συζητήσει τίποτα που έκλεισε τα χαρτιά του και τα βιβλία του πολύ θυμωμένος και είπε τέλος τη συζήτηση, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Εν πάση περιπτώσει ούτως ή άλλως η θέση του Συμβουλίου ήταν τέτοια που ε, οι πρέσβες δεν μπορούσαν να προωθήσουν πλέον τη συζήτηση, δεν είχαν δικαιοδοσία να κάνουν κάτι παραπάνω. Αυτά προτείνω λοιπόν να προχωρήσουμε σε συμφωνία πρώτης ανάγνωσης, να έχουμε τουλάχιστον κάτι, μια αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ ε, πάρα πολύ. Σας είδα στη διαπραγμάτευση ε, και είμαι σίγουρη ότι όπως και εκείνη τη φορά και όλες τις υπόλοιπες αγαπητές συνάδελφε Κάρινς δώσατε τον καλύτερο εαυτό σας. Στον κύριο Σκίνερ δίνω τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Μιλώ εξ όνος Μπέρντ Λάγκε που δεν μπορεί να παραστεί σήμερα είχατε καλέ συζητήσει μαζί του και θέλει να διαβιβάσει τις ευχαριστίες του για την εξαιρετική δουλειά και τη συνεργασία από την αρχή ω το τέλος αυτού του θέματος. Όμως ε, έχει υπάρχει ένα ζήτημα για το ότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να ανταποκριθούν σε σχέση με τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αν, έχει επενδύσει κάποιο χρόνο για τα θέματα αυτά οι σοσιαλδημοκράτες ε, θεωρούν ότι κάποια εξ ε, εξέταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να ληφθεί υπόψη για τις διεθνείς αυτές συμβάσεις ε, προτού υπογραφούν ώστε να μπορέσει πλήρως ε, να αποσαφινιστεί η συμβατότητα και το πώς συνάδουν αυτές με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καθώς αυτό λοιπόν συμπεριλαμβάνεται στα τελικά τμήματα και σε σχέση με τους συμβιβασμούς προτείνει η Σοσιαλδημοκρατική Ομάδα λέει θα προτείνει νέες τροπολογίες που θα πρέπει να ψηφιστούν όπου επιθυμεί να ενισχυθεί η νομοθεσία κατά τη διάρκεια της φάσης ε, ψήφισης προς έγκριση στην Ολομέλεια ώστε να μπορέσει αυτό το θέμα να ληφθεί υπόψη και ελπίζει ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία επ' αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βινταρκουάδρας, μετά ο κύριος Κρόισμαν. Ο κύριος Κρόισμαν, ε, θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές Έχουμε τη δυνατότητα τώρα να εγκρίνουμε το συμβιβασμό που επετέφθη και νομίζω μπορεί κανείς να το δεχθεί αυτό. Ακόμα και αν δεν πετυχαίνουμε όλα όσα θέλουμε, συμφωνούμε στο Κοινοβούλιο, όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα και θέλουμε και κάτι παραπέρα ακόμα, αλλά δεν έχει νόημα και αν μπορεί να το δεχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορεί να το δεχθεί το Συμβούλιο αυτό ως πρόταση, τουλάχιστον αυτό που έχουμε στο χέρι για την αξιολόγηση μπορούμε να το ξαναδούμε μετά από μερικά χρόνια, να εγκρίνουμε λοιπόν, εγκρίνουμε τις προτάσεις του εισηγητή. Ευχαριστώ. Άδελφος Βιντάρ Κουάδρας, ευχαριστώ πρόεδρε. Λοιπόν, ο κύριος μας εξήγησε το κείμενο του συμβιβασμού στον οποίο κατέληξε το Συμβούλιο σίγουρα κατεβάζει κάπως τις αρχικές μας ε, φιλοδοξίες γιατί θέλαμε αρκετά περισσότερα εμείς αρχικά. Θέλαμε τα ίδια τα κράτη-μέλη να μπορούν να πληροφορήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις για μια διακυβερνητική συμφωνία σε σχέση με τα ενεργειακά θέματα με μια τρίτη χώρα και αυτό να γίνεται σε σχέση με την υπογραφή προηγούμενα από την υπογραφή αυτής της συνθήκης. Στο τέλος, τέλος όμως το ε, Συμβούλιο δεν μπόρεσε να αλλάξει θέση και όλα παραμένουν τώρα στα χέρια των κρατών μελών ως αρμοδιότητα. Δηλαδή δεν θα, δεν θα συμμερίζονται τις πληροφορίες με άλλα κράτη-μέλη αν δεν επιθυμούν και μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογεί τέτοιες συμφωνίες αν το εμπλεκόμενο κράτος μέλος ζητήσει να υπάρξει μια τέτοια αξιολόγηση. Πολύ μακριά βρισκόμαστε από τις αρχικές μας επιθυμίες. Όμως έχει δίκιο ο κύριος Κάρης ότι τουλάχιστον υπάρχει υποχρέωση να κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι συμφωνίες πριν από την έναρξη σε ισχύ αυτής της συμφωνίας και εκείνες που θα προσυπογράφονται στο μέλλον όταν θα έχουν επικυρωθεί. Τουλάχιστον έτσι θα υπάρχει ένα πλαίσιο διαφάνειας και μια βάση εργασίας για το μέλλον διότι κανένας δεν απορρίπτει ιστερότερα να καταφέρουμε να πετύχουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι πολύ πιο δεσμευτικό για το Συμβούλιο. Κάπως εξεπλάγει πρέπει να πω, διότι εγώ που πολλές φορές ε, είχα ε, προεδρεύσει σε πολλούς τριμερείς ε, διαλόγους και με τον σημερινό γραμματέα αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ποτέ δεν είχα δει το Συμβούλιο να ε, έχει, ας το πω έτσι, ρίξει τα χαρτιά στο τραπέζι. Και αυτό είναι κάτι καινούριο τώρα. Και με εξέπληξε πρέπει να πω. Όμως, εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι ήταν κάτι ξεχωριστό και ε, κατεξαίρεση από πλευρά του Συμβουλίου. Συγχαίρω για την υπομονή του τον κύριο Κάνιτσο ότι πέτυχε τουλάχιστον να υπάρξει μια βάση εργασίας για το μέλλον με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ συνεργαστήκαμε στενά μαζί σου, ο κύριο Τούρμερ, και είδαμε ότι ε, βοήθησε στους ηγέτες εισηγητέ, και θα ήθελα να πω το εξή Ω πράσινη, όπως και οι σοσιαλδημοκράτε, θεωρούμε ότι αν θέλουμε η Ευρώπη να μιλά με μία φωνή, χρειαζόμαστε κάτι το οποίο να πηγαίνει ε, την παρατέρω από αυτά που έχουν συμφωνηθεί αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι επίκριση προς εσάς για τον τρόπο που κάνετε τις διαπραγματεύσεις, ε, κάθε άλλο, αλλά θέλαμε να κάνουμε μια δήλωση αντίστοιχη με τους σοσιαλδημοκράτες. Θεωρούμε ότι για να υπάρχει μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή φωνή σε αυτή τη διάσταση θα πρέπει να πάμε λίγο πέρα από αυτή τη νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Κάντινς, παρακαλώ. Σύντομα, αν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους όσους εξέφρασαν την υποστήριξή τους και τους σοσιαλδημοκράτες και τους πρασίνους που έχουν μια λίγο διαφορετική άποψη. Θα ήθελα να σας ζητήσω απλώς να σκεφτείτε τι είναι το πιο σημαντικό που έχουμε να κάνουμε εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο, στο κάτω-κάτω της γραφής. Νομίζω ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να προσαρμόσουμε την νομοθεσία και να έχουμε την καλύτερη νομοθεσία που μπορούμε να έχουμε. Η πολιτική είναι ο κόσμος του επιθυμητού που μεταφράζεται στον κόσμο του εφικτού. Και αυτό σημαίνει βάσει της νομικής βάσης ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσουν για το θέμα αυτό από κοινού. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική δήλωση. Αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν διαφέρουμε και πολύ από μια διαδήλωση στην Πλάση Λουξεμβούργ. Είναι μια πολιτική δήλωση, την ε, σημειώνουμε, αλλά δεν έχει και μεγάλη σημασία για την νομοθεσία της Ευρώπης. Ενώ εάν ε, προσαρμόσουμε αυτό το συμβιβασμό, τον εγκρίνουμε, ε, τότε έχουμε βελτιώσει τους νόμους της Ευρώπης. Είμαστε ένα βήμα, όχι όσο μεγάλο θα ήθελα εγώ να κάνω, συμφωνώ μαζί σας κύριε Τούρμες, αλλά είμαστε λίγο πιο κοντά στην κοινή ευρωπαϊκή φωνή στον τομέα της ενέργειας και νομίζω ότι εγκρίνοντας αυτή την νομοθεσία δεν θα είναι το τέλος του κοινοβουλευτικού έργου, αλλά θα είναι μόνο η αρχή. Θα μπορέσουμε στο μέλλον να την ενισχύσουμε. Και μια τελευταία παρατήρηση, σε δύο συζητήσεις που είχαμε τον Επίτροπο Έτιγκερ, και αυτό συμφώνησε ότι είναι καλύτερο να υπάρχει αυτή η συμβιβαστική νομοθεσία από το να μην υπάρχει νομοθεσία, διότι χωρίς νομοθεσία δεν είμαστε τίποτα. Και πραγματικά πρέπει να προχωρήσουμε για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο καθής μπόρεσε να εκφράσει την άποψή του και ο κύριος Κίνερ, ο οποίος δεν είναι εδώ, ε, μίλησε εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και μίλησαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Συνάδελφοι, επομένως, αύριο θα ψηφίσουμε το θέμα στην Επιτροπή. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι μπορώ να δώσω το λόγο σήμερα στον κύριο Κάλφινγκ για να κάνει μια παρέμβαση. Κανονικά η παρέμβασή του είναι για αύριο. Αύριο θα γίνει συζήτηση, διότι ε, είναι πολύ σημαντικό ο λόγο για τον οποίο πρέπει να αποσιάσει αύριο. Πρέπει να βρίσκεται στην ομάδα επαφή για τι πολιτικέ δημοσιονομικέ προοπτικέ. Μπορούμε να του δώσουμε λοιπόν το λόγο, ώστε αύριο, ακόμα και εν τη απουσία του, να μπορέσει να γίνει η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τους αγαπητούς συναδέλφους που μου επιτρέπουν αυτή την ε, αλλαγή. Δεν θα μιλήσω παραπάνω από 3-4 λεπτά και θα σας παρουσιάσω αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφορά την τροποποίηση της νομοθεσίας του 2003 για τη χρήση δημοσίων πληροφοριών. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ φιλόδοξη και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τις δημόσιες αρχές που δημοσιεύουν, απλουστεύοντας λίγο τα πάντα, ε, στο διαδίκτυο, με την εξαίρεση βέβαια προσωπικών και απόρριτων δεδομένων που είναι θέμα εθνικής ασφαλείας, ε, και επιπλέον αυτά τα δεδομένα να είναι δωρεάν ή πολύ χαμηλού κόστους. Αυτή είναι η ουσία της πρότασης και το να αλλάξουμε νοοτροπία. Δηλαδή, τα πάντα, εκτός και αν υπάρχουν κάποιοι προεριορισμοί, θα πρέπει να δημοσιεύονται. Υπάρχουν δύο βασικά επιχειρήματα υπέρ αυτή τη θέση. Το πρώτο είναι η αρχή τη δημοκρατία και της διαφάνεια τη χάραξη πολιτική και τη δυνατότητα οι πολίτε να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίε ελεύθερα από του δημόσιου φορεί. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή δημοσιεύονται αυτές οι πληροφορίες και δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν εκ νέου, θα υπάρξουν πολλές δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, ιδίω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να τις επεξεργαστούν, παρά το γεγονός ότι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εκτιμά ότι μπορεί να υπάρχουν ωφέλη της τάξης των 250 δισεκατομμυρίων ευρώ εάν χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες αυτές από επιχειρήσεις, ιδίω από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα βέβαια. Ε, συνεργαστήκαμε με τους συναδέλφους επ' αυτού, ε, ήρθαμε σε επαφή με ενδιαφερομένους, υπάρχει θέμα χρηματοδότησης. Πολλές δημόσιες αρχές πολλούν εκ νέου αυτές τις πληροφορίες και αυτό είναι τρόπος χρηματοδότηση του προπολογισμού του. Ούς έχουν ε, κάποια επιχειρήματα λοιπόν, αλλά από την άλλη ο φορολογούμενο πληρώνει τις δημόσιες αρχές για να συλλέγει και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες. Επομένως, το να τους ξαναπληρώνει δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Υπάρχει επίση μια πρόταση να δημιουργηθεί ένα εποπτικό φορέα. Αρκετέ διοικησει φοβούνται ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον γραφειοκρατικό άχθο και θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο. Υπάρχει θέμα πεδίο εφαρμογή, ποιε πληροφορίε πρέπει να δημοσιεύονται. Εδώ ισχύει η αρχή τη επικουρικότητα. Δηλαδή, κάθε κυβέρνηση αποφασίζει ποιο είναι το πεδίο εφαρμογή των πληροφοριών, αλλά βεβαίω ε, η πρόσβαση στι πληροφορίε και το δικαίωμα στι πρόσβαση στι πληροφορίε θα πρέπει να είναι ο βασικό στόχο. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν λόγοι που μας επιτρέπουν τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών. Κατόπιν, ένα χρονοδιάγραμμα. Πότε μπορούν να το κάνουν αυτό οι δημόσιες αρχές ε, και επειδή είναι δαπανηρή η διαδικασία ε, για τους νεοφερμένους, όπως για παράδειγμα δημόσιες ε, βιβλιοθήκες, ε, αρχαιοθήκες κλπ, ε, μπορεί να υπάρχει κάποιο επιπλέον κόστος. Αλλά ίσως οι μελλοντικέ πληροφορίες θα μπορούσαμε να πούμε να δημοσιεύονται οπωσδήποτε και από εκεί και πέρα όσες βρίσκονται αρχαιοθετημένες θα μπορούσαν να διατεθούν στη συνέχεια σε ψηφιακή μορφή. Και τέλος υπήρχαν και κάποιες ανησυχίες για την ανάγκη να υπάρχει ε, και ένας κατάλληλος μηχανισμός, νομίζω ότι αυτός δίνει ακριβώς τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να τις ε, πάρουν αυτές τις πληροφορίες και να τις ξαναχρησιμοποιήσουν ώστε να προσφέρουν και περισσότερες υπηρεσίες και να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα για τους πολίτες. Μπορεί να υπάρχουν λοιπόν καλές απαντήσεις στις ανησυχίες των ενδιαφερομένων και νομίζω ότι έχουμε λόγους να υποστηρίξουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πάλι να δημιουργήσουμε κάποιες νέες δυνατότητες, ε, να την πλαισιώσουμε καταλήλους, αλλά το γενικότερο σκεπτικό θα πρέπει να είναι ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι στο ε, διαθέσιμες στο διαδίκτυο χωρίς να υπάρχει ανάγκη, να υπάρχει κάποιο αίτημα. Αυτό λοιπόν ε, αφορά αυτή την νομοθεσία και πώς εγώ το προσεγγίζω. Ευχαριστώ πολύ τους κοιόδης εισηγητές από τις διάφορες ομάδες. Έχει γίνει ήδη μια συνεδρίαση ε, και ε, φαίνεται ότι θα υπάρξει και καλή συνεργασία στις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κάλφιν. Η συζήτηση για το σημείο αυτό θα γίνει αύριο. Είμαι βέβαιη ότι εάν τα καταφέρει θα είναι παρόν, αλλιώς ε, έχει αναλάβει να προασπίσει το φιλόδοξο προπολογισμό μας. Ευχαριστώ τους συντονιστές. Η συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε και ε, απλώς ευχαριστώ τους συντονιστές διότι είχαν, έδειξαν υπομονή και καθυστερήσαμε λίγα λεπτά τη συνεδρία των συντονιστών η οποία έπεται και είναι και κλεισμένο το θηρόν. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν ε, να παραμείνουν στην αίθουσα μόνο όσοι θα συμμετέχουν στη συνεδρία των συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ.